unsere erste Sitzung hier in Straßburg, oder? Ja, ja, ja. ja. I would like to start. Good morning. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Έχουμε μετάφραση α, ταυτόχρονη σε πολλές γλώσσες. Είναι η πρώτη μας συνεδρία στο Στρασβούργο αυτή δεν θα γίνουν πολλές ακόμα συνεδριάσεις στο Στρασβούργο, διότι οι συνθήκες εδώ δεν είναι ιδανικές για μας. Γιατί οι συνάδελφοι έχουν ένα σωρό πράγματα να κάνουν, να τρέχουν στη διάρκεια της ε, συνόδου. Ο συνήθω συνεδριάζουμε στι Βρυξέλλε. Εκεί είναι καλύτερε συνθήκε. Παρ' όλα αυτά όμω σα καλωσορίζω όλου θερμά. Σήμερα έχουμε στην ημέρηση διάταξη ένα σημαντικό θέμα. Οι επιπτώσεις των εγγράφων του Παναμά στις, ε, στις σχέσεις με τις αντισώμενες χώρες. Και να καλωσορίσω δύο σημαντικές προσωπικότητες που σήμερα είναι μαζί μας που έχουν σοβαρή επαγγελματική και πολιτική πείρα για να μας εξηγήσουν τα θέματα αυτά. Έχουμε καλέσει και έναν ε, δημοσιογράφο, αλλά μας έστειλε απλώς ένα μήνυμα μέσω βίντεο. Οπότε θα τον ακούσουμε στο τέλος. Και αυτοί που ήρθαν φυσικά θα είναι στην αρχή. Να χαιρετήσω λοιπόν τον Άλβεν Μοσιώμα, που είναι επικεφαλής και ιδρυτής του δικτύου για τη δικαιοσύνη για την φορολογία στην, Αφρική. Στην Ήταν επίσης επικεφαλής του συνασπισμού για τη φορολογική διαφάνεια. Είδα το βιογραφικό σας. Έχετε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο το Mainz, από την περιοχή μου. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας και περιμένουμε να μας εξηγήσετε την φορολογική πολιτική της Αφρικής γιατί είστε οι για τα θέματα αυτά. Έχετε γράψει βιβλία, δύο βιβλία για την ε, φορολόγηση και ανάπτυξη στην Αφρική μεταξύ άλλων. Καλώς ήρθατε. Να καλωσορίσω επίσης δίπλα σας τον κύριο Νούχου Ριμπάντου που είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος του Φορέα κατά της διαφθοράς στην Αφρική είναι η Επιτροπή για τα Οικονομικά και Φορολογικά Εγκλήματα. Ο κύριος Ριμπαντού ήταν επίσης επικεφαλής εισαγγελέα που συνεργαζόταν με την ε, αστυνομία της Νιγηρίας. Επίσης λοιπόν έμπειρος ε, και υπάλληλο και πολιτικός στην Αφρική για αυτά τα θέματα τα φορολογικά για τα οποία έχει παίξει θαυμάσιο ρόλο. Σας καλωσορίζουμε και εσάς ιδιαίτερα επειδή είστε και πρόεδρος της ειδική Task Force για την ε, ε, επιστροφή των εσόδων από το, πετρόλαιο, από το πετρέλαιο. Επίσης θα ακούσουμε και τον Will Fitzgibbon που είναι δημοσιογράφος που κάνει έρευνες από το, διεθνές, ε, το Διεθνή Όμιλο των Δημοσιογράφων που κάνουν έρευνες που ασχολείται ιδιαίτερα με τα έγγραφα του Παναμά. Θα οργανωθεί ως εξή η διαδικασία. Δεν έχουν έρθει ακόμη πολλοί συνάδελφοι, αλλά οι δύο συνεισηγητές είναι ε, παρόντες, οι κύριοι Κόφωτ και Γέτσεκ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Οπότε να δώσω πρώτα το λόγο σε εσά κύριε Μοσιώμα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν θα συνεχίσω όμως ε, γερμανικά. Όχι, λέει ο μπορείτε να μιλήσετε και αγγλικά-γαλλικά. Μπορώ να μιλήσω και την ε, μητρική μου γλώσσα, από όχι από ό,τι φέρετε. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας ε, τις ευχαριστίες μου στον ε, στο πάνελ σας ε, που με καλέσατε να εμένα και την οργάνωσή μου για να σας δώσω κάποιες εκ των έσω πληροφορίες για το θέμα που μας απασχολεί όλους. Εργάζομαι εδώ και 10 χρόνια για το θέμα της φορολογίας και ήταν εντυπωσιακό ότι δεν είχε δημιουργηθεί ποτέ ένας τέτοιος χώρος όπως δημιουργήθηκε με την υπόθεση των εγγράφων του Παναμά ε, για το θέμα της φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής και ιδιαίτερα σε σχέση με τον αντίκτυπο αυτής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχω μόνο 10 λεπτά, γι' αυτό θα προσπαθήσω να τα πω βιαστικά, βιαστικά και ελπίζω πως θα έχουμε το χρόνο και πάλι. Εντάξει, είναι και τόσο γεμάτη η αίθουσα, οπότε φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και για πιο συγκεκριμένα στοιχεία της δικής μου εισήγησης. Αν μπορούμε να αποκομίσουμε λοιπόν ένα δίδαγμα από τη ε, Panama Papers ε, είναι ότι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι διασυνδεδεμένη και παγκόσμιας φύσης. Οι δραστηριότητες που κρύβονται στον Παναμά έχουν άμεση επίδραση στις ζωές των ανθρώπων στην Σιέρα Λεόνε ε, οι δυνατότητες της κυβέρνησης της Ουγγάντα να παρέχει για παράδειγμα, για παράδειγμα να δίνει ε, περίθαλψη στις ε, μητέρες, να προσφέρει περίθαλψη στις μητέρες, ε, διακυβεύεται λόγω αυτής της κατάστασης και ούτω καθεξής. Όσον αφορά λοιπόν την οικονομία, είμαστε διασυνδεδεμένοι και το τι συμβαίνει σε ένα μέρος του κόσμου έχει άμεση επίδραση, άμεση επιρροή στις ζωές ανθρώπων στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Επίσης θα πρέπει να διαπιστώσουμε το παρασιτικό χαρακτήρα της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής που τροφοδοτεί σε παχυσαρκία το παγκόσμιο σύστημα το δημοσιονομικό, ε, το χρηματοπιστωτικό μάλλον. Και μόνο φωτίζοντας περισσότερο και προσφέροντας περισσότερη διαφάνεια στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αργότερα μπορούμε να συζητήσουμε και τα διαδοχικά βήματα που εμείς πιστεύουμε από τις αναπτυσσόμενες χώρες ότι πρέπει να γίνουν ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό εξ αρχής να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο το οποίο να ισχύει για όλους, αν και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το πρόβλημα της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής επηρεάζει όλες τις χώρες και όχι μόνο τις αναπτυσσόμενες. Είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει, όπως είπα, όλες τις χώρες και είναι πολύ σημαντικό να αναζητήσουμε λύσεις ε, καθολικές εξ αρχής. Και αυτό είναι για παράδειγμα εκεί που έχουμε την άμεση μας ανησυχία όσον αφορά τη διαδικασία BEPS ε, δηλαδή διάβρωση της βάσης και μετακίνησης κερδών. Ε, και τόδαμε τον αντίκτυπο αυτής της προσπάθειας, αν και προσπαθούμε μέσω περιφερειακής διαβούλευσης ε, να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή, πάντως κάποιες από τις προκλήσεις σχετίζονται με το γεγονός ότι δεν υπήρξε καθολική προσέγγιση εξ αρχής, όπως οποιοδήποτε γιατρός ε, θα σας πει ε, ότι αν έχετε εξ αρχής μια λαθασμένη διάγνωση, τότε και η αγωγή που θα σας δώσει μάλλον δεν θα είναι αποτελεσματική. Και στη χειρότερη περίπτωση μπορεί και να οδηγήσει στον θάνατο του ασθενή. Το γεγονός είναι ότι η διαφάνεια δεν μπορεί να είναι τομεακή. Και για να τα πω με τα λόγια του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ θα πω ότι η ε, αδιαφάνεια είναι ε, μια απειλή στην ε, ορθή και χρηστή λειτουργία όλων. γιατί έτσι οι εταιρείες βρίσκουν ευκαιρίες να παρακάψουν το σύστημα ενώ θα έπρεπε να έχουμε συγκεκριμένες εκθέσεις αναχώρα και να σκεφτούμε τον παγκόσμιο χαρακτήρα αυτού του φαινομένου. Ενώ αναγνωρίζουμε τον προοδευτικό ρόλο που έχει παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα εδώ το Ευρωκοινοβούλιο, καθώς ε, υποστήριξε πάντοτε μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και ε, φοροαποφυγής, ε, χρειάζεται να υπάρχει συνοχή στις πολιτικές που ασκούν και προωθούν οι μεμονωμένες οι χώρες, ώστε να μην ε, ε, δίνουμε με το ένα χέρι και το παίρνουμε πίσω με το άλλο. Γιατί αν δούμε τις συνθήκες που διαπραγματεύονται οι χώρες της Ένωσης και υπογράφουν με αναπτυσσόμενες χώρες, θα διαπιστώσουμε ότι έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ε, δυνατότητα αυτών των χωρών να, να παράγουν ε, εσωτερική, ε, εσωτερικό πλούτο για να χρηματοδοτήσουν την ίδια τους την ανάπτυξη. Περιορίζονται οι δυνατότητες αυτές μέσω των ε, συμφωνιών με τις ευρωπαϊκές χώρες και περιορίζονται και οι δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων. Τέλος, Πρόεδρε, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι δυνατότητες σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες είναι μεγάλη πρόκληση και είναι βασικό αίτιο για τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Είναι εξίσου σημαντικό να σημειώσουμε ότι δεν πρόκειται για το, πρώτο, το μόνο πρόβλημα. Η, δυνατότητα, μάλλον η δημιουργία δυνατοτήτων έχει θεωρηθεί πολλές φορές πανάκια και συχνά τάσει προ τι αναπτυσσόμενες χώρε είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε περισσότερε δυνατότητε. Υπήρξε μια μεγάλη όθηση για ένα πιο καθολικό κοινωνικό πλαίσιο, ε, να δούμε και την πρωτοβουλία για άντιση για την ε, φορολογία. Ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία για τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά δεν ήταν η μόνη και είναι σημαντικό αυτό να το έχουμε υπόψη. Αν το μόνο εργαλείο είναι, που έχεις είναι ένα σφυρί, τότε κάθε πρόβλημα μοιάζει με, με καρφί. Ε, σε αυτά έχω να, έχω να πω για την ώρα. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μοσιώμα. Τηρήσατε επακριβώς το χρόνο σας. Αυτό δείχνει ότι έχετε ζήσει στη Γερμανία. Αστεία, αστεία το είπα αυτό. Έχουμε και τις ε, γραπτές σας απαντήσεις οι οποίες ε, περιέχουν πολλή πληροφόρηση επιπλέον. Πριν λοιπόν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να δώσω το λόγο στον κύριο Νούχου Ρίμπαντου. Ευχαριστώ, θα μιλήσω αγγλικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και μέλη αυτή τη επιτροπή που με προσκαλέσατε να συμμετάσχω σε αυτή την ακρόαση. Έχω εργαστεί κατά τη διαφθοράς σε μεγάλο μέρος τη επαγγελματική μου σταδιοδρομίας, πρώτα απ' όλα ως αστυνομικός και μετά ως μέλος ε, των ανακριτών κατά της διαφθοράς και αργότερα ως πρόεδρος του πρώτου φορέα κατά της διαφθοράς στην Αφρική και στην Ε, να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε μια πολύ καλή αφορμή για την δημιουργία της ε, Επιτροπής μας που ανέκτησε 2 δισεκατομμύρια ευρώ από διαφθορά και οδήγησε πολύ κόσμο στην ε, φυλακή. Από το 2005 αλλά και μετά από την αποχώρησή μου από αυτόν τον οργανισμό μπόρεσα να μιλήσω για τον αντίκτυπο τη διαφθορά, τη λεύκανση παρανόμων προσόδων, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαπάτη. Και μπορείτε να καταλάβετε πόσο ήταν για μένα συναρπαστικό όταν ξέσπασε το σκάνδαλο των Panama Papers πέρσι. Σε ό,τι με αφορά, είναι ίσω η πιο δυνατή αποκάλυψη που είχε να κάνει με τη χρήση του εταιρικού απορρίτου, τη φοροδιαφυγή και του κρυμμένου πλούτου από τον κόσμο. Αυτή η αποκάλυψη ε, οδήγησε στην ε, παρέτηση ψηλών αξιωματούχων σε όλο τον κόσμο και ε, άρχισαν έρευνε σε πολλέ δικαιοδοσίε. Ο αντίκτυπο τη αποκάλυψη είχε μεγάλη έκταση στην Αφρική, την δική μου ήπειρο που είναι και πατρίδα μου, γιατί επί δεκαετίε οι ηγέτε και οι συνεργάτε του έχουν λαφυραγωγήσει τα δημόσια ταμεία, χωρί να του εμποδίζει κανεί. Έχουν χαθεί τουλάχιστον 50 δι δολάρια, χάνονται μάλλον κάθε χρόνο ε, σε παράτυπες οικονομικές ροές βάσει των στοιχείων του πάνελ Ταμπο για τις παράτυπες ροές από την Αφρική. Στο Πάναμα Papers εμπλέκονται πολιτικοί και ε, επιχειρηματίε από όλη την Αφρική που είχαν συνεργαστεί με τη Mossack Fonseca για να αποφύγουν το φόρο, να κρύψουν περιουσιακά στοιχεία και να πάρουν μέρο σε παραοικονομικέ συμφωνίε. Στη χώρα μου, τουλάχιστον 120 άτομα και εταιρείε εντοπίστηκαν από την εφημερίδα Premium Times που είχαν συνεργαστεί με, αυτήν την, ε, με αυτό το δικηγορικό γραφείο από τον Παναμά για να δημιουργήσουν ε, offshore εταιρείε σε φορολογικού παραδείσου. Εμπλέκονται οι πιο ισχυροί πολιτικοί τη Αφρική και οι πλουσιότεροι άνθρωποι τη Υπήρου. Βάσει των στοιχείων του Αφρικανικού Δικτύου των Ερευνητών Δημοσιογράφων Ανσύρ για το Panama Papers που καταγράφουν στοιχεία στην Αφρική, στι 52 από τι 54 χώρε τη Αφρική είχαν δημιουργηθεί offshore εταιρείε ε, με τη συνεργασία τη Mossack Fonseca η τα στοιχεία λένε ότι 44 από τις χώρες αυτές είχαν χρησιμοποιήσει τέτοιες offshore εταιρείε για να βοηθήσουν στα, να κρυφτούν τα κέρδη από ε, εμπόριο πετρελαίου, αερίου και εξόριξης, καθώς και εξαγωγών. Επίσης, ο αρχισυντάκτης τη Premium Times Μωσίκη Μοτζίντ σε μια άτυπη συζήτηση έκανε μια τεράστια αποκάλυψη. Είπε ότι οι πλουσιέτερε ε, προσωπικότητε τη Αφρική που καταγράφει το Forbes το 2016 βάσει των στοιχείων που είχαν διαρρεύσει είχαν ε, περιουσιακά στοιχεία σε όλε αυτέ τι offshore εταιρείε. Και άλλε αποκαλύψει έγιναν από του δημοσιογράφου. Για παράδειγμα, τα στοιχεία δείχνουν πόσο James Μπόρι, ένα ε, πρώην κυβερνήτη στην Ιγυρία, ο οποίος είχε υπηρετήσει πρόσφατα και ποινή κάτριξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχε ε, ακριβώς ε, συμμετάσχει σε μια τέτοια offshore εταιρεία. Και όλα αυτά χάρη στις διαρροές από τα στοιχεία σε σχέση με τη Μοσάκ Φονσέκα. Επίσης και οι μεσάζοντες σε ένα κέντρο που ε, με ε, πολλές δωροδοκίες είχε κερδίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια χάρη σε τέτοιε συμφωνίε πετρελαίου και αερίου που είχαν σχέση με την Αλγερία. Το ίδιο και ένας πρώην υπουργό πετρελαίου της Νιγηρίας που ήταν και πλουτοκράτης με ε, αεροπορική εταιρεία και πετρελαϊκή εταιρεία το ίδιο. Πάγωσαν 1,8 δισεκατομμύρια από τα περιουσιακά του στοιχεία. Το ίδιο και επιχειρηματίες. επιχειρηματίε από την Αμίμπια και ε, με συμφωνία όπλων από την Νότια Αφρική. Ε, ακόμα και από την Μοζαμβίκη ε, εντοπίστηκαν τέτοιες ε, παράνομες συμφωνίες που είχαν οδηγήσει σε μετακίνηση τεράστιους πληθυσμούς της υπαίθρου, 100.000 άτομα, προκειμένου να γίνουν συμφωνίες πετρελαίου αλλά και ένας ε, μεγιστάνας της Αιγύπτου, Σαλάχ Ντιάμπ, είχε με την εταιρεία του ε, κάνει τέτοιες ε, δουλειές. Τέλος πάντων βλέπουμε πως οι επιχειρηματίες και οι πολιτικοί ανά τον κόσμο έχουν καταφέρει χάρη στην ανωνυμία να προστατεύσουν την ιδιοκτησία τους, χάρη σε φορολογικούς παραδείσους, σε διεθνείς οργανισμούς και έχουν διατηρήσει την προτιμησιακή αυτή ιδιοκτησία το πάνελ της Αφρικανικής Ένωσης καταγράφει τις παράνομες οικονομικές ροές από εταιρείε και ζητά την συνολική παγκόσμια δράση για να καταπολεμηθούν οι φορολογική παράδοση, η παράδειση ανά τον κόσμο. Χρειάζεται συντονισμένη διεθνής δράση για να καταπολεμηθούν οι φορολογική παράδοση και ε, δικαιοδοσίε που προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα χρηματοοικονομικού απορρίτου. Ο πρόεδρο του πάνελ της Αφρικανική Ένωσης και πρόεδρο τη Νοτιοαφρική Τάμον Μπέκη ε, ζήτησε να δοθεί τέλος σε αυτό το σύστημα. Επίσης, ψηφίστηκε ένα σύστημα για να σταματήσει η προτιμησιακή διοκτησία εταιριών πρόσφατα ε, στην Νιγηρία σε μία, μάλλον ο πρόεδρος Μουχαμάντου Μπουχάρη της Νιγηρίας σε μία ε, σύνοδο στο Λονδίνο κατά της διαφθοράς εξέφρασε τη δέσμευση της κυβέρνησής του να σταματήσει προτιμησιακή ε, ιδιοκτησία εταιριών στην χώρα του. Το ίδιο και στην Κάνα πέρασε ένα σχετικό νόμο για τι εταιρείε και την προτιμησιακή ιδιοκτησία το Δεκέμβριο του 2016. Σε ένα ε, σεμινάριο δύο ημερών στην Άκρα το Φεβρουάριο, οι οργανισμοί ε, Πρωτοβουλία Κεραιότητα τη Γκάνα, ε, Διεθνή Διαφάνεια και Κέντρο Προάσπισης των Πολιτών, αλλά και άλλες οργανώσει από την Κένια και το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τις ε, προκλήσεις σε σχέση με την προτιμησιακή ιδιοκτησία και την απόκρυψή του. Ε, η Γκάνα, η Κένια και η Νιγηρία αποφάσισαν να δημιουργήσουν από κοινού ένα νομικό σύστημα που να συγκεντρώνει τα στοιχεία τη ιδιοκτησία των εταιριών και να καταπολεμά το απόρριτο. Δείχνει η περίπτωση του Πάναμα Papers την ανάγκη να καταπολεμηθεί η διαφθορά διεθνώ και να έχουμε ένα διαφανέστερο κόσμο. Καλό τι αφρικανικέ κυβερνήσεις και όσους έχουν παραβιάσει τον νόμο να φροντίσουν να τους διώξουν και να εντοπίσουν αυτές τις εταιρείες offshore. Χρειάζονται ακόμα πάρα πολλές έρευνες, αλλά χρειάζεται και η δική μας πυγμή για να υπάρξει δίωξη. Σας ευχαριστώ για τη δράση που θα αναλάβετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ριμπαντού. Δεν ανέφερα, αλλά ήσασταν ο επικεφαλής εισαγγελέας με την Ιγυριανή αστυνομία και σας διόρισε και σας διόρισαν τα Ηνωμένα Έθνη και επικεφαλής ε, της ομάδας ε, επιτήρησης στο Αφγανιστάν το 2011. Σημαντικές ε, λοιπόν αρμοδιότητες. Έχουμε εδώ τον δημοσιογράφο, ο οποίος θα μας έστειλε ένα μήνυμα μέσω βίντεο, αλλά νομίζω ότι καλύτερα να τον ακούσουμε στο τέλος. Το κείμενο της ομιλίας του δημοσιογράφου είναι ήδη διανεμημένο Οπότε τα επιχειρήματα, τα επιπλέον που αναφέρονται, μπορείτε να τα διαβάσετε. Και αν στο τέλος δεν προλάβουμε να δείξουμε το βίντεο, θα σας στείλουμε το link για το βίντεο. Εντάξει, αυτή θα ήταν η πρότασή μου. Αν συμφωνείτε, να συνεχίσουμε και καταρχάς να ευχαριστήσω τους δύο μιλητές άλλη μια φορά λοιπόν για την εισαγωγή τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ποιες είναι οι διαστάσεις του προβλήματος στην Αφρική. 52 αφρικανικές χώρες ε, αναφέρονται στα έγγραφα του Παναμά και είχε παρέμβαση η Μοσάκ Φονσέκα σε 44 από αυτές. Είπατε ότι το BEPS ε είναι ένα θέμα ΟΣΑ και ευρωπαϊκό που δεν πρέπει να το ξεχάσουμε σε σχέση με την Αφρική. Οπότε προτείνω Έχουμε εδώ το κατάλογο μιλητών και θα ξεκινούσα με τον ε, Γέπε Κόφορτ και τον Πίτερ Γέτσεκ που είναι οι δύο συνεισηγητές μας. Γέπε και έχεις το λόγο. Πέντε λεπτά ε, να είναι το κάθε, η κάθε διαδικασία. Ένα λεπτό ερώτηση, τέσσερα λεπτά απάντηση. Ευχαριστώ για την παρουσία σας, λέει ο κύριος ε, βλέπουμε τι επιπτώσεις έχει η φοροδιαφυγή και η αποφυγή στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τρομερή, οι υπολογισμοί της Oxfam σε 52 αναπτυσσόμενες χώρες θεωρεί ότι θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί 269 δισεκατομμύρια για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και να υπάρξει ανάπτυξη αν είχε υπάρξει σοβαρή καταπολέμηση της φοροδιαφυγή. Είναι πολύ περισσότερο από την αναπτυξιακή βοήθεια που δίνουμε στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Πολύ σημαντικό λοιπόν. Επίσης, η υπόθεση Μοσάκ Φονσέκα είναι μόνο σταγόνα στον ωκεανό. Είναι μια εταιρεία δικηγόρων στον Παναμά αυτή. Αλλά υπάρχουν πολλές άλλες εταιρείε που δεν έχει αποκαλυφθεί ο ρόλο του. Αναφερθήκατε η διαφάνεια. Είπατε ότι είναι κλειδί. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω. Εμείς ε, κάνουμε πολλά. Έχουμε την υποβολή εκθέσεων αναχώρα από τις πολυεθνικές. Τι περισσότερα θα μπορούσαμε να κάνουμε στην νομοθεσία μας για να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να επιτύχουν περισσότερη διαφάνεια. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια πρόταση για τις εκθέσεις αναχώρα αλλά αυτή ε, δεν περιέχει τα στοιχεία αναχώρα. Είναι απλώς συνολικά τα στοιχεία για όλες τις αντισωμένες χώρες. Επίσης υπάρχει πρωτοβουλία για τον πραγματικό δικαιούχο. Τι μπορούμε να κάνουμε, Να υπάρχει ίσως ε, ένα παγκόσμιο μητρό για τους πραγματικούς δικαιούχους. και για τους φορολογικούς παραδείσους. Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να τηρούν. Μετά υπάρχει ένα διαδικαστικό θέμα. Ε, υπάρχουν κοινέ προδιαγραφέ για την υποβολή εκθέσεων, αλλά οι αναπτυσσόμενε χώρε ε, δεν έχουν την αναγκαία διοικητική ικανότητα για να συμμορφωθούν με αυτά τα πρότυπα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Παρακαλώ και οι δύο ομιλητέ θα μπορούσαν να απαντήσουν. Ποιο θέλει να αρχίσει. Ευχαριστώ. Καταρχάς, ε, ποια είναι η γνώμη μας για το ποια είναι τα βασικά θέματα για τη διαδικασία BEPS. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, η διαδικασία δεν μας περιέλαβε από την αρχή. Αυτό που παρατηρούμε στην ε, συνεχιζόμενη διαβούλευση είναι ότι θα εφαρμοστεί διαφορετικά η διαδικασία BEPS ε ε, ανάλογα με τις χώρες και τις περιφέρειες. Για τις χώρες της Αφρικής, για παράδειγμα. Κυρίως ασχολείται με τις ε, πρώτες ύλες. Και αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο BEPS. Κάθε φορά που τίθεται θέματα αυτά, είναι ότι δεν μπορούμε να σας παράσουμε στοιχεία που δεν είναι μέσα σε αυτά που έχουν καθοριστεί. Δεν μπορούμε δηλαδή να συζητήσουμε τα ουσιαστικά θέματα γιατί δεν είναι στο πεδίο αναφοράς. Το ίδιο για τα φορολογικά κίνητρα. Το εξετάζουμε εδώ και πολλά χρόνια, εγώ και άλλοι συνάδελφοι. Πώς δηλαδή διαβρώνεται η φορολογική βάση από τον αθέμητο φορολογικό ανταγωνισμό. Μπορείτε να, μπορεί να γνωρίζετε ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες προτιμούν την φορολόγηση στην πηγή. Ενώ στις ευρωπαϊκές χώρες ε, προτιμούν την φορολόγηση με βάση τον τόπο κατοικίας ή την έδρα των επιχειρήσεων. Όπως είπατε, Πρέπει να γνωρίζετε λοιπόν γιατί πολλέ αναπτυσσόμενε χώρε ο καθορισμός ε, των τιμών μεταφοράς είναι πολύ δύσκολος. Το είπε και ο Νούρου προηγουμένω. Δεν έχουμε ούτε καν μονάδες για την μέτρηση των τιμών μεταφοράς. Οι διαδικασίε λοιπόν ε, αυτόματης ανταλλαγής προφοριών αμοιβαία θα μας βοηθούσαν. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε στην πράξη επιτόπου σε κάθε αναπτυσσόμενη χώρα ε, τις απαιτήσει αυτές. Πώς θα σας στείλουμε τα στοιχεία όταν δεν έχουμε καν την έννοια του πώς υπολογίζονται οι τιμές μεταφορών. Η τιμολόγηση ε, μεταφορών. Στην Ιγυρία, ξέρετε, ένα μεγάλο τμήμα του προπολογισμού μας ε, είναι από τις πρώτες ύλες που πουλάμε. Άρα η φορολόγηση παίζει μικρότερο ρόλο. Και κάτι ακόμη. Στην ουσία, Το θέμα είναι να συμμετέχουν όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες στο καθορισμό αυτών των διαδικασιών. Αλλά πρέπει να το δούμε και από την πλευρά το πώς επηρεάζει την καθημερινότητα των χωρών. Να συνεχίσω σε αυτό που είπε ο συνάδελφος. Το πιο σημαντικό που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να παίξει ηγετικό ρόλο να, να ψηφίζει σωστούς νόμους για να τους ε, αντιγράφουν οι άλλοι. Εάν υπάρχει ένα σημαντικός ε, πολιτικός συνασπισμός που να παίρνει μια πολύ σωστή και διαφανή θέση, τότε αυτό περνάει και αλλού, διαδίδεται στις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου. Οι υπόλοιπες χώρες απλώς εφαρμόζουν αυτά που και εσείς έχετε επιτυχώς κάνει. Ένας νόμος από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να έχει μεγάλη επίπτωση και σε άλλα μέρη του κόσμου γιατί θα παίξει έναν εκπαιδευτικό ρόλο. Θα δείξει και σε άλλους πώς να αντιμετωπίσουν τα κοινά προβλήματα. Οπότε αυτό θέλουμε να σας πούμε. Παίξτε πρωτοπόρο ρόλο. Να αναλάβετε πρωτοβουλία και να είστε φυσικά δίκαιοι και έναντι των μικρών χωρών που δεν έχουν την ικανότητα και την τεχνογνωσία για να κάνουν τα πράγματα όπως εσείς. Εδώ μπορείτε να επιτύχετε πολλά. Αλλά πρέπει να γίνει σύντομα. Γιατί τώρα είναι η στιγμή, τώρα υπάρχει μια κινητικότητα. Ας μην επιτρέψουμε να χαθεί η ευκαιρία. Επίσης πρέπει να βοηθήσετε τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες να αλλάξουν την νομοθεσία τους. Για παράδειγμα, να έρθετε σε επαφή μαζί τους. Να καταλάβουν τι κάνετε εσεί. Θα τι βοηθήσετε να καταλάβουν τι πρέπει να γίνει. Τρίτον, αυτό που είπατε κι εσείς. Ορισμένες ε, ορισμένες ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτούς που ε, κλέβουν τους πόρους μας και τους πάνε εκεί που δεν μπορούμε πια να τους ανακτήσουμε. Πρόκειται για τους φορολογικούς παραδείσους. Εάν υπάρχει τρόπος να ε, καταργήσετε τους φορολογικούς παραδείσους, να το εξετάσετε. Βεβαίως, μπορείτε να μας βοηθήσετε, μπορείτε να ε, εκπαιδεύσετε τις φορολογικές μας αρχές, τις αρχές επιβολής του νόμου, τα μέσα. Σας ευχαρίστησα για τη βοήθεια που δώσατε στην Επιτροπή μας για την καταπολέμηση του φορολογικού και οικονομικού εγκλήματος το 2005. Μας δώσατε 24 εκατομμύρια δολάρια. Και ως ε, συνέπεια ανακτήσαμε πάνω από 24 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω της εργασία μας. Και έχουμε επιτύχει την καταδίκη σε φυλάκιση άνω των 500 ατόμων. Χάρη σε αυτή τη βοήθεια που μα δώσατε. Να πώ μπορείτε να μα βοηθήσετε λοιπόν διάφορες προτάσεις και να διευκολύνεται την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω απλούστευσης των διαδικασιών. Να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά που έχετε. Μόνο μέσω αυτής της συνεργασίας θα μπορέσουμε να πιάσουμε τους κακούς στον κόσμο. Γκέτσεκ και μετά οι πολιτικές ομάδες. Αλλά πρώτα απ' όλα λοιπόν ο συνεισηγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε για την παρουσία σας. εκτιμάται ιδιαίτερως και για τις παρουσίες σας. Θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε από τη δική σας οπτική γωνία το άλλο τμήμα της ε, όλης αλυσίδας. Δηλαδή οι οικονομικές ροές πάνε κάποιες φορές και από την Αφρική προς την Ευρώπη σε μια πρώτη φάση. Ξέρετε σε ποιες χώρες της Ευρώπης υπάρχουν ε, ιδιαίτεροι δεσμοί κάποιων αφρικανικών χωρών με ευρωπαϊκές. Κάποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν περισσότερο παράνομο χρήμα από ό,τι άλλες. Και υπ' αυτήν την έννοια, την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την ε, επιβολή της, πώς τη βλέπετε, μπορεί να βελτιωθεί και στον κατάλογο των χωρών υψηλού κινδύνου που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό επεξεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούν να δοθούν κίνητρα σε αφρικανικές χώρες για να τακτοποιήσουν κάπως την οικονομική τους αυτή κατάσταση και τις οικονομικές τους σχέσεις. Ωραία, ποιος θα ξεκινήσει τώρα τις πολιτικές ομάδες, παρακαλώ. να αναφερθώ στην έκθεση που ανέφερε και ο Νούχο. Την έκθεση του πάνελ υψηλού επίπεδου. Αυτό που αναφέρει είναι ότι πέραν το γνωστό ποσό των 50 δις που χάνουν ετησίως αυτές οι χώρες εξηγεί ότι είναι δύσκολο για τις παράτυπες οικονομικές ροές να εντοπίσουν εντοπίσουμε τους φορολογικού σε ανά τον κόσμο. Είναι στην Καραϊβική, είναι στην Ευρώπη, υπάρχουν και στην Αφρική. Ο δικό μου οργανισμός, όπως ε, συζητάμε αυτή τη στιγμή, προσπαθεί να εντοπίσει στην Κένια έναν ακόμη φορολογικό παράδεισο μέσω ενός διεθνούς κέντρου που λειτουργεί εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ακόμα και στις αναπτυσσόμενες χώρες να υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Θα σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει κανένα σοβαρό σκάνδαλο διαφθοράς στην Ήπειρό μας, θα το διαβεβαιώσω και ο Νούχου, που να μην έχει σχέση με κάποιο φορολογικό παράδεισο. Όλα τα όλα τα οικονομικά σκάνδαλα θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε τα, τα νησιά Κέιμαν, ο Παναμάς, Εδώ το διεθνές σύστημα πρέπει κάτι να προβλέψει. Και τι θα μπορούσε να γίνει. Εμείς από την Αφρική αντλούμε κάποια θετικά διδάγματα για το τι ρόλο μπορούν να διδραματίσουν οι βουλευτές. Εάν ειδικά το Ευρωκοινοβούλιο δεν είχε δώσει τέτοια προβολή στην δουλειά του πάνελ μας, δεν θα είχαμε καταφέρει να πετύχουμε τίποτα σε παγκόσμια κλίμακα. Κοιτάζουμε λοιπόν τι μπορούμε να μάθουμε από την Αφρική. Πρόσφατα δημιουργήθηκε ένα βουλευτικό φόρουμ, κοινοβουλευτικό φόρουμ για τι πράτυπε οικονομικέ ροέ που προσπαθεί να φέρει μαζί οι βουλευτέ από όλη την Ήπειρο για να δούμε πώ μπορούμε να προβάλλουμε και να εκθέσουμε τα θέματα αυτά. Διότι οι λύσει πρέπει να προκύψουν και σε εγχώριο επίπεδο δηλαδή τους φορολογικούς δασμούς, τις φορολογικές μάλλον συμφωνίες που υπογράφουν ε, οι χώρες μας, τα συγκεκριμένα όρια που προβλεπόνται για τους φορολογικούς δασμούς, συμφωνίες με φορολογικούς παραδείσους, και σίγουρα ανάμειξη των βουλευτών, των κοινοβουλίων. Αυτό είναι ε, ε, μια σημαντική διάσταση για πολλές αρχές είναι καθοριστική σημασία η ενημέρωση και για τις εφορίες, τους φορολογικές, τους αρχές, τις αρχές κατά της διαφθοράς. Τα όρια όμως που έχουν προβλεφθεί για να μπορέσει κανείς να έχει πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες είναι τόσο ψηλά που γίνονται απαγορευτικά για ορισμένε αναπτυσσόμενε χώρες. Πρέπει λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι τα όρια, λόγω χάρη για τη διαδικασία υποβολής έκθεσης αναχώρα, να μην είναι εξαιρετικά αυστηρά. Πολλέ χώρε στην Αφρική έχουν χαμηλό ΑΕΦ, οπότε εάν δείτε τι έγινε με το Panama Papers, έχουν τέτοια όρια που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα στοιχεία, όπως έγινε με το Panama Papers. Ευχαριστώ. Ναι, εσείς. Ναι, εάν υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επίσης ε, σχετίζονται με το βρώμικο χρήμα. Τώρα όχι. Πριν από 10-15 χρόνια ναι. Όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε στο πάνελ μας, είχαμε κάποιες περιπτώσεις που ερευνήσαμε. Την περίπτωση της Αμπάντζα, του Αμπάντζα, ε, ο οποίος από την Ιγυρία έκλεψε 6 δις δολάρια και τα πήγε βόλτα ανά τον κόσμο. Ένα μέρος ήταν στην Ελβετία. 1,2 πέρασαν από τις Βρετανικές αρχές. Όμω τα πράγματα αλλάξαν από τότε που ξεκινήσαμε τι έρευνε. Είχαμε δυσκολίε με κάποιε χώρε, αλλά τελικά μα στήριξαν. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο λόγου χάρη μα στήριξε πολύ και καταφέραμε να έχουμε αποτελέσματα. Καταφέραμε μάλιστα στην περίπτωση του Αμπάντζα να πάρουμε και πίσω και κάποια δις δολάρια από τον ελβετικό του λογαριασμό θυμάμαι ότι τότε είχα γράψει σε δικαστικούς λειτουργούς στη Γαλλία για να ζητήσω βοήθεια και φανταστείτε ότι επειδή έγραψα στα αγγλικά τους πριν δύο χρόνια να το μεταφράσουν στα γαλλικά αυτό που είχα γράψει. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω ε, και δεν ξέρω αν είναι εδώ η κυρία Ζολή, κυρία Εύα Ζολή. Τι, φοβερή γυναίκα είναι αυτή. Τι εξαιρετική γυναίκα που καταλαβαίνει το πρόβλημα του αναπτυσσόμενου κόσμου. Ε, πραγματικά έκανε ό,τι μπορούσε ε, προκειμένου να μας βοηθήσει και είμαστε πολύ περήφανοι για το αποτέλεσμα. Ελπίζω να μην σας φέρνω σε δύσκολη θέση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσω ανθρώπους όπως η Ευαζόλη που πραγματικά μας βοήθησαν στην προσπάθειά μας. Τώρα έχουν αλλάξει βέβαια όλα. δεν συμμετέχουν πολλές χώρες ε, στην ε, τήρηση τέτοιων λογαριασμών πέρα από το Λευτεριστέα και κάτι άλλες μικρές. Εκτός Ευρώπης γίνονται συνήθως αυτές οι δουλειές. Αλλά έχετε όλοι χρήμα. Μπορείτε να κάνετε κάτι για αυτές τις περιπτώσεις. Αν τους ασκήσετε πίεση, μπορεί να σταματήσει αυτή η συμπεριφορά. Σας διαβεβαιώ δεν υπάρχει καθαρό χρήμα στους φορολογικούς παραδείσους. Δεν έχει κανείς καμία δικαιολογία για να διατηρεί χρήμα σε φορολογικούς παραδείσους. Ούτε ουδε μια. Ε, είναι για λόγους εγωιστικούς και προσωπικούς συμφέροντος και μυστήριους βρώμικους που τηρεί κανείς, διατηρεί δηλογαριασμούς σε φορολογικούς παραδείσους. Δεν έχει κανείς λόγο εάν έχει κερδίσει νόμιμα τα χρήματα του να τα πάει στη Μαδέρα ή οπουδήποτε αλλού. Ε, εάν έχει ένα νόμιμο εργοστάσιο που λειτουργεί κανονικά λόγω χάρη. Ε, φτάνει πια, αυτό έχουμε να πούμε, όπου και αν είναι αυτό το χρήμα στον κόσμο και ελπίζουμε στη βοήθεια όλων σας. Ευχαριστώ. Ε, επέτρεψα οι απαντήσεις να είναι λίγο πιο αναλυτικές και γι' αυτό θα ήθελα, επειδή έχουμε περιορισμένο χρόνο τώρα που θα μιλήσω προς των ομάδων, να είστε λίγο πιο ε, συνθετικοί για να προλάβουμε. Ο κύριος Τόμ Φαντε Λάρε. Σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να απευθύνω την ερώτησή μου στον κύριο Μουσιούμα. Όπως είπε ο κύριος Τριμπάντα, οι αφρικανικές χώρες χάνουν δεκάδες ε, ε, εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, καθές οι πολυεθνικές ε, φοροδιαφεύγουν. Αυτό επικυρώνεται από ένα σωρό εκθέσεις που γνωρίζουμε και αυτές οι δραστηριότητες όχι μόνο εμποδίζουν την ανάπτυξη των χωρών σας, αλλά αποτελούν και παγκόσμιο πρόβλημα καθώς οι παράνομες ροές φτάνουν σε τρομοκρατικές ομάδες όπως η Μπόκο Χαράμ ή η Αλ Σαμπάμπα. Ο κύριε Μουσίμα, όταν μιλήσατε για περισσότερη συνοχή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή στις πολιτικές που εμείς χαράζουμε, η ερώτησή μου είναι ποιο ρόλο βλέπετε να μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της φοροδιαφυγής στην Αφρική. Μπορείτε αυτό να το αναπτύξετε περισσότερο και έπειτα όταν μιλήσατε για οικοδόμηση δυνατοτήτων. Η αλλαγή στην οτροπία καταρχάς πρέπει να προέλθει λέτε από τις ενδιαφερόμενε χώρε στην Αφρική ή από την Ένωση και του διεθνεί οργανισμού όπω ο ΣΑ ή ο ΙΕ που μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο. Ποιο πρέπει πρώτο να κινηθεί κατά τη γνώμη σα. Και μια τρίτη και τελευταία ερώτηση που έχω είναι έχετε διαπιστώσει ειλικρινέ ενδιαφέρον από οποιαδήποτε αφρικανική χώρα για να λύσει το πρόβλημα τη φοροδιαφυγής. Δηλαδή, αν έπρεπε να κάνετε ποιοι είναι οι καλύτεροι μαθητές, να κάνετε κατάλογο των καλύτερων μαθητών Ποιοι είναι αυτοί, οι πρώτοι τρεις στην Αφρική. Πώς θα απαντήσει πρώτος, παρακαλώ εσείς. Ε, αποφασίστε μεταξύ σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Για το θέμα της ε, συνέπειας και της συνοχής της πολιτικής. Θα ήθελα αυτό να το συγκεκριμενοποιήσω και να το θέσω στο πλαίσιο της φοροδιαφυγής. Κάθε φορολογικός παράδεισος πουλάει κάτι ιδιαίτερο. Προσπαθεί να καθοριστεί, ε, λες και έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι πάλι στην Ευρώπη, για παράδειγμα, αν και έχουν καταβληθεί προσπάθειες για να γίνουν ε, έλεγχη για το ποιες είναι οι επιρροές ε, των συμφωνιών που κάνουμε εμείς ε, με τις αφρικανικές χώρες. Παρ' όλα αυτά υπάρχει διάχυση, υπάρχει αντίκτυπος, υπάρχει... Θα πρέπει να γίνει πιστεύω αναχώρα αλλά και μια πανευρωπαϊκή ανάλυση του είδους των, συμφωνιών που συνάπτονται με τους οικονομικούς εταίρους της Αφρικής. Δεν βλέπω γιατί να μην μπορεί να γίνει μια πιο συνολική ανάλυση για το πιο είναι ο γιατί αυτό που θα συμβεί και αυτό ε, ε, βασίζεται σε παρελθούσα εμπειρία ε, κάποια στιγμή που ε, εγώ είχα επαφές με ε, υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών της Ολλανδίας και της Βρετανίας και είπαν ναι, θα επανεξετάσουμε τις συμφωνίες που υπογράψαμε με το Μαλάουι. Αλλά φυσικά αν το Μαλάουι έχει υπογράψει κακή σύμβαση με το Ηνωμένο Βασίλειο, εμείς θα υπογράψουμε μια καλύτερη. Ε, πρέπει δηλαδή καθένα να μπορεί να προστατεύει το συμφέρον του. Δηλαδή να μην ορίζεται το, το, το όριο από το ποια συμφωνία έγραψε το Μαλάουι με το Ηνωμένο Βασίλειο μόνο. Αυτό προς τα κάτω μας τραβάει, ενώ μια πιο συνολική ανάλυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να ενθαρρύνει ε, μια ευγενή άμυλα προς τα πάνω. Τώρα, δεν υπάρχει μόνο μία λύση. Ε, θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες ε, σε εθνικό επίπεδο και διάφορες κυβερνήσεις έχουν κάνει πρόοδο. Όσον αφορά τις φορολογικές συμβάσεις υπάρχουν συμφέροντα. Η Κένια διαπραγματεύεται με το Μαουρίσιος. Θα φανταζόταν κανείς ότι οι πλούσιοι μαυρικιανοί το προωθούν, εν, αλλά στην πραγματικότητα οι κενιάτες επιχειρηματίες θέλουν να χρησιμοποιήσουν το μαυρίκιο για να επενδύσουν. Μπορεί κανείς να διερωτηθεί πώς αυτό το τόσο μικρό νησί είναι ο μικρότερος, είναι ο μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων ε, για την Ινδία, ας πούμε. Ινδικέ επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τον μαύρο και έτσι, δηλαδή ω φορολογικό παράδεισο. Εμείς λοιπόν θέλουμε να πιέσουμε τις ίδιες μας τις κυβερνήσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το είδος τα προ... συμπεριφορές. Τώρα, ποιοι είναι οι καλοί μαθητές. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Αυτό που βλέπουμε είναι δύο βήματα μπροστά, ένα βήμα πίσω γίνονται συνήθως. κάνει κάποια προοδευτικά βήματα μια χώρα και μετά ξαναπίσω. Στην Κένια, ας πούμε, μετά μια μεγάλη όθηση, όπου η χώρα έβαλε, θέσπισε τον νόμο Θάμπο ε, αλλά μετά άλλαξε το καθεστώς, ε, συγκεντρώθηκαν οι επιχειρηματίες, ε, πίεσαν την καινούργια, την καινούργια κυβέρνηση. Στη Ζάμπια το ίδιο. Είχαμε μια κυβέρνηση που αύξησε τη φορολογία στον εξωτερικό τομέα, άλλαξε το καθεστώς και ό,τι είχε φτιαχτεί και πήγε πίσω. Οπότε η κοινωνία των πολιτών ό,τι κάνει, ξανά αρχίζει τη διαδικασία, πιέζει τους ξένους επενδυτές να ζητήσουν, να απαιτήσουν κτλ χώρες όπως η Κένια, η Γκάνα, η Νότιος Αφρική έχουν παίξει σημαντικό ρόλο όχι μόνο ε, στηρίζοντας και ενισχύοντας τις δυνατότητές τους τις ίδιες αλλά και ε, προσπαθώντας να δουν πώς μπορούν να μεταφέρουν αυτές τις δυνατότητες σε χώρες της περιοχής τους υπό την Αφρικανική ε, Συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να στηρίξει λύσεις λοιπόν επιτόπου. Η δημιουργία δυνατοτήτων μπορεί να γίνει εντός της Αφρικής. Η Νότιος Αφρική, Α πούμε, μπορεί να τις μεταφέρει τις εμπειρίες της στις υπόλοιπε χώρες της περιοχής της και η Κένια το ίδιο. Συγγνώμη, Πρόεδρε, που μακρηγόρησα. Μια ακόμα παρατήρηση από τον κύριο Λεμπάντο. Ναι, σύντομο θα είμαι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που λείπει στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ο τρόπος που παρουσιάζουμε αυτά που θέλουμε. Μεγάλοι σε ομάδες, μπλοκ όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να μας στηρίξουν οικονομικά. Δηλαδή να στηρίξουν αυτό που θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις δυνατότητές μας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα με τι, τι κάνει η Διεθνής, ε, υπηρεσία, ε, Διεθνής Αναπτυξιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασίλειου. Έχει επενδύσει πολύ σοβαρά ε, για να εντοπίσει πού μπορεί να βάλει λεφτά και να έχει αποτελέσματα. Το τμήμα κατά της διαφθοράς λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Έχουν δαπανίσει εκατομμύρια και εκατομμυρίων. Και οι φορολογικές τους αρχές λειτουργούν πολύ καλύτερα και αυτό έχει κάνει τεράστια διαφορά. Μπορείς να πας σε όλες αυτές τις χώρες και να δεις τι θα, τι θα, πού τα χρήματα σου θα δώσουν αποτέλεσμα. Έχει να κάνει με τα χρήματα και επίσης μέσα από όλα αυτά μπορείτε να τα μας μάθετε πώς θα διαχειριστούμε αυτούς τους πόρους πιο καλά και πιο αποτελεσματικά. Εάν υπάρχει ο, τρόπο, τρόπος να δαπανηθούν σωστά τα χρήματα και να έχουμε αποτέλεσμα κάθε φορά. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι ε, θέμα πόρων, είναι θέμα ε, άμεσης δέσμευσης, να, άμεσης όμως ε, δέσμευσης και δαπάνης των χρημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τώρα 8 ομιλητές από τις ομάδες και 4 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ σήμερα, διότι μπορεί να ξέρετε ότι το 2015 το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα, το οποίο ζητούσε από την Επιτροπή με ένα πρόγραμμα δράσης 10 σημείων να υποστηρίξει τι αναψώμενες χώρες για να καταπολεμήσουν τη και φοροαποφυγή. Εγώ ήμουν μεταξύ των εισηγητών ε, του ψηφίσματο και πραγματικά βρίσκω όλα αυτά που περιείχε να αντικατοπτρίζονται στη σημερινή συζήτηση. Πολύ σύντομα λοιπόν πρώτο σημείο τότε ζητούσαμε να αυξηθεί το κομμάτι της αναπτυξιακής βοήθειας που στηρίζει αυτές τις δραστηριότητες. Ξέρετε συνάδελφοι ότι ήταν το 1% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας το 2011 αυτό που αφιερώνονταν σε αυτούς τους σκοπούς. Προφανώς δεν έφτανε. Έπειτα ζητούμε οι κυβερνητικοί φορείς σε επίπεδο Αφρικανικής Ένωσης να αναλάβουν ε, ρόλο. Μόνο έτσι μπορούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να συμμετάσχουν ισότιμα στη συζήτηση για τη διευθέτηση των θεμάτων αυτών. Συνάδελφοι, αυτά έπρεπε να συζητηθούν και στην Αντισαβέμπα, ε, ε, όπως και γίνει μάλλον στην Αντισαβέμπα και πρέπει να ξαναγίνει. Να ξαναγίνει φέτος στο σχετικό φόρουμ και οι ε, αναπτυσσόμενες χώρες να πιέσουν και άλλο για ένα διαφερνητικό φόρουμ. Για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, με συγχωρείτε πρόεδρε για τα κρόνημα, προσπαθώ να συντομεύσω. Νομίζετε ότι μια μεταβατική περίοδος ίσως να ήταν τρόπος για να αποφύγουμε την αμοιβαιότητα που αποκλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες και για την υποβολή ε, εκθέσεων αναχώρα. Μιλήσατε για τα όρια προκειμένου να έχει πρόσβαση κανεί στα δεδομένα, όμω για τι φορολογικέ συμφωνίε. Θεωρείτε ότι πρέπει να ε, πιέσουμε περισσότερο ώστε να έχουμε φορολογικέ συμβάσει μέσω του ΟΗΕ και όχι μέσω του ΟΣΕ και φορολογικέ συμφωνίες και για την διαφάνεια σε σχέση με την προτιμησιακή ιδιοκτησία. Υπάρχουν περιφερειακά πλαίσια όπως προσπαθούμε να κάνουμε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα δικό μας πλαίσιο, υπάρχει μόνο εθνική συζήτηση για εθνικές καταγραφές και μητρώα. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάζω και το ρολόι μου πλέον. Παρακαλώ. Ναι, πολλές ερωτήσεις και λίγος χρόνος. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απολύτως για σας για την ανάγκη ενός διεθνούς φορέας στην αιγύδα του ΟΗΕ για τα Σίγουρα υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία του όσα, αλλά σίγουρα όσα ε, θεμητό είναι να προωθεί τα συμφερόντα των χωρών του όσα. Εκεί πρέπει να γίνει ένα βήμα πρόοδου και νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί αποφασιστικά τουλάχιστον από την πλευρά της να στηρίξει αυτή την πρόθεση. ώστε να υπάρξει ένα περιθώριο και οι αναπτυσσόμενε χώρε να συμμετάσχουν στη συζήτηση των θεμάτων αυτών για την προτιμησιακή διοκτησία. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα για πολλές αναπτυσσόμενε χώρες, όμως δεν μπορούμε να το δούμε σε γεωγραφικά στεγανά. Πρέπει να υπάρξει διεθνή συντονισμό σε πολλέ χώρε τη Αφρική. Νιγηρία, Κένια, Νοτιοαφρική, Ναμίμπια που έχουν δεσμευτεί για εθνικό μητρό, αυτό είναι κάτι, αλλά τι κάνει αυτό τελικά μακροπρόθεσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, βοηθάει να υπάρξει καλύτερο σχεδιασμό για πολλά πράγματα, αλλά για την επιμέρους φορολόγηση, unitary taxation, θυμάμαι τι είχε γίνει πριν από 5-6 χρόνια που είχαμε συζητήσει κάτι ανάλογο. Και η αντίδραση ήταν ακριβώ η ίδια. Οι ε, εκθέσει αναχώρα δεν είναι πρακτικέ, δεν είναι αποτελεσματικέ. Έχουν βελτιωθεί, υπάρχουν περισσότερε λεπτομέρειε, υπάρχουν περισσότερε πληροφορίε και αποδεκτικά στοιχεία. Αυτό δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πιέσει προ τη σωστή κατεύθυνση όταν θέλει. Αλλά ο ρόλος που μπορούν να παίξουν οι επιμέρους γεωγραφικές περιοχές, όπως στην περίπτωση του Unitary Taxation, ας πούμε, της ε, επιμέρους φορολόγησης, είναι περιορισμένος. Πρέπει να δούμε πιο σφαιρικά τα θέματα για να μπορούμε να υπολογίσουμε και τον αντίκτυπο στι αναπτυσσόμενε χώρε. Ε, θα ήθελα να πω περισσότερα, αλλά με πιέζει ο πρόεδρο. Ευχαριστούμε κύριε Ριμπάντη. Ε, ναι, σε συνέχεια όσον είπε. Συμφωνώ απολύτω και τα υπογραμμίζω και εγώ. Αλλά αυτό που είπατε η ανάγκη να αυξήσετε την απτυξιακή σας βοήθεια. Είναι κρίσιμη σημασία. Να καταλάβετε ότι ο καλύτερο τρόπο να βοηθήσετε τι αναπτυσσόμενε χώρε είναι να έχουμε εμεί τι δυνατότητε. Εμεί να μπορούμε να δώσουμε απάντηση στα φορολογικά, με φορολογικέ αρχέ και δικέ μα δυνατότητε να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά. Εάν αυτά τα δύο γίνουν, σε πέντε χρόνια σα διαβεβαιώ, δεν θα βλέπετε πια κανέναν Αφρικανό μετανάστη στην Ευρώπη πρέπει να φροντίσουμε με τους πόρους που έχουμε να κάνουμε ε, ό,τι καλύτερο μπορούμε. Με ένα καθήκον να οικοδομήσουμε καλό οικοδευτικό σύστημα, να φτιάξουμε δρόμους, να έχουμε καλή στέγαση. Αν τα είχαμε όλα αυτά στις χώρες μας δεν θα φεύγαμε. Κλαίμε καθημερινά όταν βλέπουμε τους νέους να εγκαταλείπουν την Ήπειρο. Θέλουν μια καλύτερη ζωή. Δεν μπορούμε να τους δώσουμε επιτόπου. Αυτό θα μπορούσατε να κάνετε, να καταλάβετε πώς μπορούν να κάνουν περισσότερα, να χρησιμοποιήσουν αυτά που έχουν, να σταματήσει αυτή η σπατάλη. Εάν στις αφρικανικές χώρες δινόταν αυτή η ευκαιρία, θα μπορούσαν όλοι να φροντίσουν τους εαυτούς τους. Παρακαλούμε, βοηθήστε. Βοηθήστε με τη βοήθεια και τους πόρους. Μην πετάτε τα λεφτά σας στα θέματα της μετανάστευσης. Τώρα δώστε τα. Επενδύστε και ε, δώστε χρήμα αβέρτα τα επόμενα πέντε χρόνια για αυτά τα θέματα. Θα δείτε σε πέντε χρόνια ότι θα συζητάμε στι επιτροπέ για τη μετανάστευση. Πρέπει να φανούμε έξυπνοι εδώ. Εσεί να φανείτε έξυπνοι και να σκεφτείτε διορατικά το μέλλον. Πόρου για να μπορούμε εμεί να φροντίσουμε του εαυτού μα. Είναι και άλλα τα ζητήματα μεν, αλλά Ευχαριστώ πολύ. Ήταν έκκληση προς εμάς να δούμε ριζική αλλαγή για αυτά που κάνουμε και πέρα από τα αφρολογικά θέματα. Επόμενος, Πύρκο Ρούινεν Λέρνερ από το ECA. Πύρκο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για όλη αυτή τη χρήσιμη πληροφόρηση που ακούσαμε σήμερα το πρωί. Έχω μια ερώτηση που έχει να κάνει με την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ρόλο που παίζουν στην ρύθμιση του, της παγκόσμιας ε, φορολογίας. Τι μπορούμε να κάνουμε. Σε πολλές χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου παίζει μεγάλο ρόλο πώς μπορούν να λάβουν δάνεια. Το 2015 η Παγκόσμια Τράπεζα είπε ότι θέλει οι χώρες αυτές να κάνουν περισσότερα για να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή. Δεν ξέρουμε όμως τι έχει επιτευχθεί επί τόπου. Γιατί υπάρχουν και μια σειρά από άλλα στοιχεία. Τι μπορούμε να κάνουμε για να παίξουν και οι ίδιες αναπτυσσόμενες χώρες πιο, πιο ε, αποφασιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Ποιος θα ξεκινήσει, παρακαλώ εσείς. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Συμφωνώ ότι η Παγκόσμια Τράπεζα και το Δέλτα ΝΙΤΑΦ έχουν κεντρικό ρόλο και όντως συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις σε επίπεδο των χωρών μας για τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Σε πολλές χώρες γίνονται προσπάθειες μεταρρύθμισης και ενίσχυσης ε, των δυνατοτήτων των ε, φορολογικών αρχών και μεταρρύθμιση της νομοθεσίας και από τη χώρα μου. Με πολύ μεγάλη βοήθεια από αυτούς τους δύο οργανισμούς. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει ανταγωνισμός με αυτούς τους δύο οργανισμούς για τα φορολογικά κίνδρα για παράδειγμα μας έχουν πει πως ε, δεν είναι χρήσιμα αυτά τα μέσα για να προσελκύσουμε ξένες ε, απευθείας επενδύσεις, άμεσες επενδύσεις. Αλλά από την άλλη μεριά οι ίδιοι οργανισμοί κάνουν, ε, εκπονούν και ορισμένα μητρώα για την φορολογική ελκυστικότητα κάποιων χωρών, κάτι το οποίο δείχνει ότι έχει σημασία ο φορολογικός ανταγωνισμός για να προσελκύσει κανείς ξένες επενδύσεις. Πολλές χώρες στην Αφρική και όχι μόνο στην Αφρική αλλά και αλλού στον αναπτυσσόμενο κόσμο χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα ανισοτήτων. Αλλά η Παγκόσμια Τράπεζα μας λέει θεωρεί ότι μπορείτε να συλλέγετε με τρόπο ε, που να μειώνετε... Ε, όσο ε, ανέρχεται το εισόδημα και κατόπιν να διανύμεις προς τους φτωχότερους και μας ε, πιέζουν να εισαγάγουμε τον ΦΠΑ για παράδειγμα. Μας λένε πρώτα να συλλέξετε πόρους με τον ΦΠΑ και μετά να δείτε πώς θα διανύμετε αυτούς τους πόρους. Αλλά αυτό μας δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Γιατί θεωρούμε ότι έτσι θα αυξήσουμε τις ανισότητες του φορολογικού μας συστήματος. Δηλαδή θα επιβαρύνουμε περισσότερο τους φτωχούς. Και υπάρχει μεγάλη αντίσταση σε χώρες όπως η Γκάνα, η Σιέρα Λεόνε. Οι πολίτες είναι κατά και ανθίστανται στην ε, εισαγωγή του ΦΠΑ, όπω και στη χώρα μου την Κένια. Διότι βεβαίως έτσι διευκολύνεται η συλλογή φόρων. Λαμβάνουμε λοιπόν αντικρουόμενα μηνύματα από τους οργανισμούς αυτούς για το τι πρέπει να κάνουμε ως αναπτυσσόμενες χώρες. Ναι γενικά η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι οργανισμοί μας έχουν βοηθήσει πολύ, με εκπλήσουν ορισμένα που ακούω. Είναι, είναι πραγματικά ε, ε, πηγή γνώσης που μας βοηθάει. Ίσως θα έπρεπε να μας βοηθήσουν περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα τα ξέρουν όλα αυτά. 150 χρόνια ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ε, ξέρουν πολύ καλά πώς να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουν τεράστια γνώση. Για παράδειγμα για τα φορολογικά καθεστώτα. Χρηματοδότησαν την μηχανογράφηση της ε, υπηρεσίας μας στη χώρα μου. Λαμβάνουμε πολύ βοήθεια λοιπόν από την ε, Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ Εντάξει, μπορεί κάποιε συμβουλέ που μα δίνουν να μην είναι οι καλύτερε, αλλά αν θέλετε να αναπτύξουν τη δυνατότητά του κάποιε χώρε, τότε πρέπει κυρίω να βασιστείτε σε αυτού του δύο οργανισμού. Είναι πολύ καλή η συνεργασία μαζί του, αν θέλουμε οτιδήποτε στον τομέα μα να επιτευχθεί. Ευχαριστώ, Λουί Μισελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που προσκαλέσατε τους δύο εμπειρογνώμονες από την Αφρική Νομίζω ότι έχουμε ένα κοινό αγώνα να κάνουμε για το θέμα αυτό. Και είμαι όλο και πιο πεπισμένος αγαπητοί συνάδελφοι ότι πρέπει να έχουμε έναν ε, ριζικά διαφορετικό στρατηγικό πολιτικό ε, στόχο. Δεν νομίζω ότι με μικρομεταβολές ε, διαφορετικέ πολιτικές θα επιτύχουμε τίποτα. Μπορεί να μην έχω ριζοσπαστική νοοτροπία, αλλά εδώ πρέπει να είμαστε ριζικοί. Πρέπει να εργαστούμε σε ένα παγκόσμιο δεσμευτικό πλαίσιο. Αν κάνουμε μικροαλλαγές δεξιά-αριστερά πάνω και κάτω, δεν θα επιτύχουμε τίποτα. Επίσης θα πρότεινα κύριε Πρόεδρε η Επιτροπή μας να στείλει μια επιστολή στους διοργανωτές της ε, συνάντησης κορυφής Αφρικής Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αμπιτζάν τον Νοέμβριο για να θέσουν αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μου ανέθεσε να προετοιμάσω τις διαπραγματεύσεις μετά το Κοτονού και θα φροντίσω να είναι αυτό το θέμα στη μέση διάταξη. Έτσι θεωρώ ότι θα προωθήσουμε το τόσο σημαντικό αυτό θέμα. Θα σας εκπλήξει το ότι δεν θα εξαντλήσω τα δύο λεπτά μου, αλλά ήθελα να κάνω αυτή την πρόταση. Επαναλαμβάνω. Με μικροαλλαγές δεν θα επιτύχουμε τίποτα. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι, πολύ πιο ακραίοι. Εγώ είμαι μετροπαθής και με ενοχλεί, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να είναι κανείς ακραίος. Νομίζω ότι αναπτύσσεται όλο και πιο πολύ η οικονομία της αγοράς στην Αφρική και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, ακόμη πιο σημαντικό, να υπάρξει κάπως σοβαρή φορολογική πλαισίωση του. Ευχαριστώ πολύ. Τι σχόλιο έχετε. Δεν υπήρχε ερώτηση. Οπότε ένα σύντομο σχόλιο. Συμφωνώ. Οπωσδήποτε πρέπει να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην Αφρική και τι μπορούμε να στηρίξουμε. Οι αφρικανικές φορολογικές αρχές κάνουν ε, τρομερές προσπάθειες για να αναπτύξουν το δυναμικό. Πρέπει να έχουμε τέτοια προγράμματα τα οποία θα συνδυαστούν με αυτά που κάνουμε επιτόπου. Έτσι δημιουργήσαμε αυτό το consortium με επικεφαλής τον ε, Τάμπο που προσπαθούν να συνδυάσουν τις προσπάθειες σε εθνικά και περιφερειακά επίπεδα για να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή. Η βοήθεια που μπορεί να δώσει η Ένωση είναι ακριβώς να στηρίξει αυτά που ήδη γίνονται. Άρα ήδη δηλαδή θα βοηθήσει κάτι που είναι ήδη εγκινήσει. Και εγώ συμφωνώ. Και όπως είπατε βεβαίως πολλές αλλαγές λαμβάνουν χώρα στην Αφρική. Νομίζω ότι έχουμε καλύτερους ηγέτες σήμερα που θέλουν πραγματικά να υπάρξουν βελτιώσεις και αλλαγή. Ορισμένοι λοιπόν έχουν μάθει και είναι διατεθειμένοι να μάθουν από αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΩΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα. Έχουμε λοιπόν αυτή την ειδική ομάδα. Έχουμε τις πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών. Όλα αυτά σιγά σιγά συγκεντρώνονται και έχουν τεράστια επίπτωση. Και δεν βλέπω να ανθίσταται κανείς από τις αφρικανικές χώρες στην προσπάθεια βελτίωσης. Είναι μια ευκαιρία που πρέπει να την αδράξουμε. Και σας διαβεβαιώ και παγκοσμίω αυτή είναι η λύση όπως είπατε. Η Αφρική είναι έτοιμη για οποιαδήποτε στήριξη και βοήθεια μπορεί να λάβει από οπουδήποτε. Ευχαριστούμε. Ο Ματ Κάθη για την ΚΟΥ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. και ε, εξαιρετικέ παρουσιάσει και ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα το πρωί. Ήθελα απλώ να θέσω και εγώ κάποιε ερωτήσει σε σχέση με τον αντίκτυπο των Αφρολικών Συμφωνιών για την ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών ιδίω τη ρήτρα κατά της κατάχρησης και υπεξέλιξης. Και αν έχετε τα σχετικά στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον ΝΟΣΑ και για το πόσο οι εμπορικές σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να περιλαμβάνουν μια τέτοια ρήτρα κατά της, εξέρ, της κατάχρησης ή υπεξαίρεσης. Εδώ λοιπόν χρειάζονται σχετικές διευθετήσεις. Έχετε κάποια ιδέα λοιπόν για το κατά πόσο αυτή η ρήτρα θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική φορολογικής φορολογικές συμφωνίες. Έχετε κάποια θέση για το τι θα μπορούσε να επιτευχθεί. Και μια δεύτερη ερώτηση για την ε, ανάλυση over ε, Αναφέρατε την ε, υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Έχετε κάποια άποψη για το τι ρόλο μπορεί να παίξει η υποβολή εκθέσεων αναχώρα και να επηρεάσει την ανάλυση μας συνολικότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Εσείς, ξεκινήστε. Συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω οι συστάσεις με τη ρήτρα υπεξαίρεσης θα ε, περιόριζαν ιδιαίτερα στον αρνητικό αντίκτυπο των δυσμενών ιδίως φορολογικών συμφωνιών. Είδαμε οι αναπτυσσόμενες χώρες να υπολείπονται πολύ των προτεραιοτήτων ε, των όσων θα έπρεπε να συμβαίνουν. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν χώρες που έχουν προβλέψει μορατόριουμ για φορολογικές συμφωνίες. Η Κένια, λόγου χάρη, εξαιτία ιδίω του Panama Papers. Διότι υπήρχε μια εταιρεία πατρελαίου και εξορρυκτική, η οποία εκτέθηκε, αποκαλύφθηκε μέσω του Panama Papers ότι είχε προσπαθήσει να δίνει όσο λιγότερο φόρο μπορούσε στις φορολογικές αρχές. Μοροτόριο, λοιπόν από την Κένια. Και καταγγείλαμε την ε, συμφωνία από τον οργανισμό μας, από το φορέα μας, καταγγείλαμε τη συμφωνία της Κένιας με το Μαυρίκιο. Το ίδιο και στην ε, Ζάμπια, την Γκάνα. Αυτό δείχνει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει και το Κοινοβουλίο σας και η Ευρωπαϊκή Ένωση. για να έχουμε μία ρήτρα κατά, της κατάχρησης. Η θεμελιώδης αρχή πάντως της υποβολής έκθεσης χώρα είναι να δούμε κατά πόσον μπορεί να είναι δημόσιες και να ισχύουν και όλες τις χώρες. Έτσι δηλαδή φαίνεται να δημιουργείται ένα υβριδικό σύστημα. Και θα έπρεπε να φροντίσουμε να έχουμε μια συνολικότερη εικόνα τώρα για τα όρια. Πρέπει να φροντίσουμε να ε, γίνει σωστή προσαρμογή για να μπορούν και οι αναπτυσσόμενες χώρες να, να από την όλη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος για τους πρασίνους, Judith Sargentini. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε, κύριοι, είσαστε πολύ ευγενικοί μας. Γεμίσατε φιλοφρονήσεις και μας ε, ζητήσατε να είμαστε ένα παράδειγμα για την Αφρική και τον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ. Εδώ Να κάνουμε όμω μια διάκριση μεταξύ φορολογικών ε, παραπτωμάτων που είναι απλώ αδικήματα ή ε, τη διευκόλυνση τη φοροδιαφυγή και φοραπάτη. Εμεί ακόμα διευκολύνουμε, διευκολύνουμε τι δικέ σα εταιρείε και τι δικέ μα πολυεθνικέ να παίρνουν τα κέρδη από τι δικέ σα τι χώρε και να τα φέρουν εδώ για να πληρώσουν λιγότερο φόρο. Είμαι συνεισηγήτρια για τι διαπραγματεύσει τη οδηγία περί τη καταπολέμηση του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο και το βλέπουμε το θέμα αυτό με 28 κράτη-μέλη που δεν θέλουν την διαφάνεια τελικά για τους πραγματικούς προτιμησιακούς ιδιοκτήτες, ιδίως όταν πρόκειται για καταπιστεύματα ή άλλου είδους χρηματοοικονομικούς ε, σχηματισμούς. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, πέραν των ποινικών αδικημάτων, και για όσα βλέπετε σε σχέση με τη φοροδιαφυγή εκτός Αφρικής, όπου χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά συστήματα, που δεν είναι μόνο ε, ηθικά, μόνο νομικά, αλλά και ηθικά προβληματικά κάποια φορά. Τι θα μπορούσε να γίνει. Ναι, το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που θέσατε αυτό το ερώτημα. Η διαφορά μεταξύ διαφυγής και αποφυγής είναι το ύψος του τείχους της φυλακής. Στην μια περίπτωση πάντα φυλακή, στην άλλη όχι. Στις... Από την οπτική γωνία των αναπτυσσόμενων χωρών βεβαίως κάνει διαφορά. Εάν το χρήμα το, απόσ... το απέσπασε κανείς με παράνομα ή νόμιμα μέσα. Και για να ξαναέρθω στο θέμα των δυνατοτήτων. Γιατί να θέλει μια εταιρεία να φοροδιαφεύγει όταν μπορεί να φοροδιαφύγει νομίμως. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια ενίσχυσης των ε, συστημάτων στην πράξη. Μιλήσαμε για τις τιμές μεταβίβασης, το transfer pricing. Και πρέπει να δούμε και τις δυσκολίες ανάπτυξης που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας σε σχέση με τους ανθρώπινους πόρους, τους συγκρίσιμους δείκτες. Πρέπει να αναζητήσουμε στοιχεία που να αντικατοπτρίζονται στο σύστημα όπως θα λειτουργεί. Όπως και η όλη διευθέτηση του ΟΗΕ με την ομάδα κρούσης που προσπαθεί να ε, καταρτήσει τη σωστή μεθοδολογία για την καταπολέμηση των παράτυπων οικονομικών ροών. Εδώ αυτό που βλέπουμε με τη γυναίκα είναι ότι η υποβολή εκθέσεων αναχώρα Προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται στην περίπτωση της εταιρεία. Τι κάνουν, απλώς παίρνουν το κέρδος τους, και το πάνε αλλού, ε, αποφεύγουν το φόρο. Δηλαδή πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που θολώνει το τοπίο και δεν μπορούμε να δούμε πραγματικά την ε, δραστηριότητα της κάθε εταιρεία. Είναι μια αρχή το σύστημα υποβολής εκθέσεων ανά χώρα. Ναι, τα ίδια μας απασχολούν και εμάς. Παρακαλώ. Ναι, εγώ μια δήλωση πολιτική, όχι φοροτεχνική όπως ο συνάδελφος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει τεράστια διαφορά για τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, αρκεί να έχει κανείς την τόλμη να ε, υψώσει τον και να κάνει το σωστό. Η διαφάνεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κάτι το κακό, ούτε η λογοδοσία. Η αντίσταση στους νόμους δεν είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσει κανείς. Θυμάμαι όταν η Αμερική προσπαθούσε να περάσει τον ανάλογο νόμο για τη διαφθορά που ε, ότι όλες οι πολυεθνικές εταιρείες είναι υπόλογες για την ε, κακή διαχείριση εκτό ΗΠΑ. Ήταν αντιδημοφιλή ο νόμο αυτό, αλλά η Αμερική θεώρησε ότι θα βοηθήσει να κάνει καλύτερε business η Αμερική γενικότερα στο μέλλον. Και τελικά έτσι αποδείχθηκε. Όλοι εμεί που είμαστε στην πρώτη γραμμή του πολέμου κατά τη διαφθορά, αν βλέπουμε ότι τις καλύτερες πρακτικές τις έχουν τελικά οι αμερικανικές εταιρείες γιατί έχουν ε, νόμο που τις αναγκάζει να είναι υπόλογες με μια ε, πετρελαϊκή εταιρεία στην ε, Νιγηρία που ερευνήθηκε λόγω χάρη να σα διαβεβαιώσω ότι δεν είχε ανάμειξη καμία αμερικανική εταιρεία λόγω του νόμου τους. Και όποτε υπήρξε διαγωνισμό για κάποια σύμβαση, οι αμερικανικέ εταιρείε είχαν ε, συγκριτικό πλεονέκτημα, διότι είχαν την νομοθεσία τη δική του, την εγχώρια, και απέφευγαν την ε, κακή διαχείριση ή συμπεριφορά. Γι' αυτό σας λέω να έχετε την τόλμη και να προχωρήσετε. Δεν θα χάσετε τίποτα. Καμία εταιρεία δεν θα τα πάει άσχημα λόγω της λογοδοσία ή της διαφάνειας. Και αν μιλάμε για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαφάνεια. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί τίμοι και δίκαιοι για όσα κάνουμε. Έτσι θα αλλάξετε το τοπίο για τις αναπτυσσόμενες χώρες με νόμους που τις κάνουν να λογοδοτούν, να είναι διαφανείς. Ό,τι και να κάνει κανείς μπορεί να ε, προασπιστεί τις εταιρείε όπου και αν λειτουργούν στον κόσμο. Δεν θα το μετανιώσετε ποτέ. Ευχαριστούμε από τον EFTD ε ο κύριος Κόμπα. Thank you very much. We are now... Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Πολύ, πολύ, κύριοι, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μα είπατε. Αλλά βεβαίω οι αναπτυσσόμενε χώρε βεβαίω και χρειάζονται του φόρου. Αλλά πολλοί φοβούνται ότι θα, τα χρήματα που θα βάλουν στην άκρη θα του τα βουτήξει το κράτος, οι γγκάντε. Ή όλοι μαζί αυτοί. κυβερνήσεις, οι γκαγκστερ Η ιδιωτικότητα στι ε, στις είναι σημαντική. Εμείς εδώ το έχουμε συνηθίσει, αλλά στι αναπτυσσόμενε χώρες ε, φοβούνται επίσης ε, μήπω κάποιο του πιάσει όμοιρους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχει κάνει τον ιδιωτικό του ε, χώρο και αυτό έχει χρησιμοποιηθεί ως χώρος για να αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει, να παρέμβει σε διάφορα θέματα φορολογικά και επιχειρηματικά. Όμω ειλικρινά δεν είναι δική μα υπόθεση. Κατά τη γνώμη μου κάτι τέτοιο θα είχε νεοπικιακό χαρακτήρα. Τα αφρικανικά έθνη θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα προβλήματά τους και να λάβουν τις ευθύνες για τις δίκαιες τους εταιρείες και να προχωρήσουν προς τον ελεύθερη επιχειρηματικότητα και τον καπιταλισμό. Εγώ έχω περισσότερη εμπιστοσύνη στις χώρες αυτές της Αφρικής. Ε, και μην φορτωθείτε με ένα σωρό κανονισμούς που εμποδίζουν τις εταιρείες ε, όπως στην Ευρώπη ή στην Αμερική και αλλού. Γιατί η έλλειψη κανονισμών βοηθά την Αφρική να ανταγωνιστεί και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα και δεν πρέπει να αφήσετε το, εδώ αυτούς τους ανθρώπους να σας το πάρουν. Και Ναι, δύο λεπτά έχετε μιλήσει. Βάλτε την ερώτησή σας. Συμφωνείτε μαζί μου πως ίσως Υπάρχει κίνδυνος να χάσετε την ανταγωνιστικότητά σας και ίσως αυτό να είναι ένας ε, ε, δούριος ύπος που προσπαθούν να σας πουλήσουν οι εδώ. Μάλιστα. Για να μην χρειάζεται να μου φωνάξει ο πρόεδρος και να μου κλεισβεί στο μικρόφωνο, θα προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημά σας, χρησιμοποιώντας ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα. Εγώ ζω στο δεύτερο όροφο στο σπίτι μου. Στο τρίτο όροφο Διαπιστώνω, μάλλον, και διαπιστώνω ότι έρχεται υγρασία και σχηματίζονται λεκέδες στο ταβάνι μου. Ο λόγος είναι γιατί από τον τρίτο όροφο υπάρχει διαρροή και μάλιστα η διαρροή ήταν πίσω από το κρεβάτι του τρίχρονου παιδιού της από πάνω οικογένειας. Κάλεσα λοιπόν τον, ε, τον γείτονα, του είπα κοίταξε είναι ένα νοικιασμένο αυτό εδώ το σπίτι, δεν είναι δικό μου πρόβλημα, στο δικό μου χώρο όλα είναι καλά. Αφόσον έχεις πρόβλημα εσύ, μίλα με το δικό σου ιδιοκτήτη γιατί είναι στο δικό σου ταβάνι το πρόβλημα και όχι στο δικό μου πάτωμα. Για εκείνον όλα ήταν εντάξει. Η κουζίνα του ήταν εντάξει, το πάτωμά του ήταν εντάξει. Προσπάθησα λοιπόν να το αντιμετωπίσω, δεν έγινε τίποτα. Λίγου μήνε αργότερα ε, προκλήθηκε μια ρογμή λόγω αυτής της υγρασίας και χρειάστηκε εκείνος να μετακομίσει. Γιατί σας λέω αυτό το παράδειγμα. Γιατί η υπόθεση που κάνετε ε, ότι οι αφρικανικές χώρες θα πρέπει μόνο τους να λύσουν τα προβλήματα είναι λανθασμένη. Γιατί όπως αποδείχτηκε από τα Panama Papers, τα, οι πόροι που βγαίνουν από την Αφρική δεν πηγαίνουν στην Αφρική, αποθηκεύονται κάπου αλλού κρύβονται κάπου αλλού όλα αυτά τα χρήματα, εκατομμύρια εκατομμυρίων, δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων και δεν τα παίρνουν μέσω με βαλίτσες, αλλά μέσω, περνάνε μέσω αξιοσέβαστων ευρωπαϊκών τραπεζών. Γι' αυτό μπορεί κάτι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις να δουν τι μπορούν να κάνουν γιατί αυτό επηρεάζει όχι μόνο τους άλλους από την άλλη πλευρά αλλά έχει επιπτώσεις και στις δικές τους οικονομίες και τους ε, πολίτες σύντομα να πω και εγώ ότι σήμερα ο κόσμος είναι παγκοσμιοποιημένος. Αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Παγκοσμιοποίηση υπάρχει, ό,τι και αν γίνεται κάπου επηρεάζει και όλους τους υπόλοιπους. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και όποιος ε, προσπαθεί να τα αλλάξει αυτά χάνει το χρόνο του. Είναι θέμα χρόνου να συνειδητοποιήσει όλος ο κόσμος ε, ότι αυτό ισχύει. Κοιτάξτε, δεν ξέρω από πού είστε. Είστε μάλλον από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μα εσεί είσαστε στην Ιγυρία 100 χρόνια. Εσεί μα ε, απικήσατε. Δεν μπορείτε να έρχεστε και να μα λέτε ότι δεν έχετε φέρτε καμιά ευθύνη για το τι συμβαίνει σήμερα στην Ιγυρία. Είναι, είναι αμέτρητοι οι πόροι που φύγαν από την Ιγυρία και πήγαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και πρέπει να καταλάβετε ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι. Είμαστε ένα και το αυτό. Αν λέτε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση νύπτουμε τα σχήρες μας και και, και, βγάλετε τα πέρα μόνοι σας. Μα πω γιατί ήρθατε τότε στην Ιγυρία, σας κάλεσε κανείς τότε. Ευχαριστώ για αυτήν την ε, έκκληση που έγινε με τόσο πάθος. Δεν ήταν μόνο το Ενωμένο Βασίλειο απικιακή δύναμη, ήταν και άλλες. Δεν μπορώ να επιτρέψω συμπληρωματικές ερωτήσεις. Έχω την Μπάρμπαρα Κάπελ και τον Φρανκ Έγγελ και μετά τέσσερις διαδικασίες προσέλκυσης της προσοχής του Πρόεδρου. Η Μπάρμπαρα πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ είμαι από την Αυστρία. Όπως ξέρετε, εμείς ε, δεν υπήρξαμε απικιακή δύναμη. Οπότε δεν έχω πρόβλημα με όλα αυτά. Θέλω να σε ευχαριστήσω όχι μόνο γιατί ήρθατε σήμερα εδώ, αλλά γιατί είχαμε μια πολύ ζωηρή συζήτηση με έντονα συναισθήματα για το θέμα αυτό, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που από μόνο του μπορεί να φαίνεται βαρετό. Και θεωρώ ότι επιβεβαιώσατε κάτι που συχνά το ακούμε, ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής χρειάζεται παγκόσμια αντιμετώπιση. Ακούγεται ωραία, αλλά είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Γι' αυτό οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες του ΟΣΑ, των Ηνωμένων Εθνών και μας είπατε ότι για τις αναπτυσσόμενες χώρες θα ήταν ε, σημαντικό να υπάρξουν πρωτοβουλίες του ΟΗΕ. Ξέρω και από τα κείμενα ότι ακριβώς ο φόρος ε, επί των κερδών των επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντικός γιατί στις χώρες σας ε, τουλάχιστον το 25% των πόρων προέρχεται από αυτό το φόρο. Αν δεν έχετε αυτούς τους πόρους δεν έχετε χρήματα για την υγεία, για την παιδεία, για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Και είναι ακριβώς αυτό που είπατε κύριε Ριμπαντού. Εάν δεν έχετε τους αναγκαίους πόρους, τότε φεύγουν οι άνθρωποι. Και αυτό είναι άσχημο και για εκείνους και ούτε για μας είναι καλό. Θεωρώ λοιπόν ότι και εγώ δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω μαζί σας, πρέπει να σας βοηθήσουμε να μας βοηθήσετε. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Και μετά είπατε δύο πολύ σημαντικά ότι πρέπει να ενισχυθούν οι πόροι που δίδονται από την αναπτυξιακή βοήθεια για να αναπτύξετε τις δυνατότητες της ε, χώρας σας και των υπηρεσιών σας για να ανακτηθούν οι πόροι, για να πληρώνουν οι επιχειρήσεις πόρους και ότι χρειαζόμαστε περισσότερε συμφωνίε εμπορίου και φορολογική συνεργασία, γιατί πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε δεν έχουν επαρκή συμφωνίε με τι ε, χώρε τη Ένωση. Και αυτό σημαντικό δίδαγμα. Ναι, ναι. Τρει ερωτήσει. Τι μπορείτε να κάνετε εσεί, Πρέπει να κάνουμε και εμεί αυτά που πρέπει να κάνουμε. Υπάρχουν μια σειρά από πρωτοβουλίε σε, ε, αφρικανικό επίπεδο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Μία είναι η Επιτροπή για τις Φορολογικές Υποθέσεις και η Πλατφόρμα για την Φορολογική Συνεργασία που δημιουργήθηκαν για να ληφθούν μέτρα ανάπτυ... Ε, στήριξης των αναπτυσσόμενων χωρών στον τομέα της φοροδιαφυγής. Πώς προχωράει η εφαρμογή των μέτρων αυτών. Δεύτερη ερώτηση. Λέτε δεν σας βοηθάει το BEPS. Γι' αυτό είχατε την άλλη αυτή πρωτοβουλία, ATIF, και επίσης για την Ιγυρία. Υπάρχει σύσταση του ΟΣΑ. Ε, πώς έχει εφαρμοστεί αυτή η σύσταση. Ε, είπα δύο, ήταν τρία. Το, πότε μας μένουν δύο λεπτά για τις απαντήσεις. Δύο λεπτά για τις απαντήσεις σας, παρακαλώ. Όχι ο καθένας. Δύο λεπτά και δύο μαζί. Θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσω σε ένα λεπτό τόσο σημαντικά θέματα. Σύμφωνο. υπάρχει ουσιώδης ανάγκη ενίσχυσης ε, των δυνατοτήτων των εφοριακών μας αρχών. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε ξανά και ξανά. Στην Τανζανία, για παράδειγμα, πριν από δύο μήνες, δημιουργήθηκε μια ειδική, τιμή για τις, ειδική μονάδα για τις τιμές μεταβίβασης. Και μέσα σε λίγους μήνες είπαν ότι από τρεις πολυεθνικές ε, μπόρεσαν να ανακτήσουν 200 εκατομμύρια. Παράλληλα έχουμε τέτοια παραδείγματα στην Ουγκάντα με καλά αποτελέσματα. Ναι, λοιπόν, η ανάπτυξη των διοικητικών δυνατοτήτων είναι πολύ σημαντική. Αλλά δεν είναι πανάκια. Πρέπει να δούμε ευρύτερα το θέμα. Πώς να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο πλαίσιο που να τους περιλαμβάνει όλους. Και εδώ μπορεί να βοηθήσει ο ΟΗΕ. Ευχαριστώ για τη στήριξή σα Πέντε δευτερόλεπτα ακόμη, λέει πρόεδρος. Ναι. Η Νιγηρία εφαρμόζει κατά γράμμα όλες τις υποδείξεις του ΟΣΑ και όλων των άλλων ε, θεσμών που μας ε, βοηθάνε. Και ε, το φορολογικό μας καθεστώς είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με άλλες χώρες και όχι μόνο η Νιγηρία. Οι περισσότερες αφρικανικές χώρες είναι διατεθειμένες να μάθουν είναι ανοιχτές. Ορισμένες φορές απλώς δεν έχουμε την τεχνογνωσία. Το πώς θα το κάνουμε ακριβώς. Αυτό είναι η πρόκληση. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ που, διατηρήσατε το, που τηρήσατε το χρόνο σας. Και μετά τον Φρανκ Έγκελ, τέσσερις για, την, για το Catch the Eye. Ναι, θα είμαι σύντομος. Το καλό με τον να από το Λουξεμβούργο δεν αντιμετωπίζεται ποτέ ω απεικιοκράτη είναι πολύ μικρός και αδύναμος για να θεωρηθεί κακός απεικιοκράτης. Τέλος παντών, είπαμε πάρα πολλά για τα ύποπτα χρήματα και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εκεί δεν είμαστε τόσο άσπηλοι. Ε, έχω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο μόνη στην Ήπειρο. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε και να βοηθήσουμε, αλλά υπάρχουν και άλλοι και νέοι φορείς στην Ήπειρο σα. Η Κίνα, η Τουρκία, η Ινδία, η Βραζιλία σε κάποιο βαθμό με τις πορτογαλόφωνες χώρες. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ως προς τις ευαισθησίες αυτών των φορέων και σε σχέση με όσα μόλις συζητήσαμε και τα προβλήματα αυτά, τις δυσκολίες αυτές. Ποιες είναι οι διαφορές πώς βλέπετε την, ε, την ε, στάση των ε, μελλοντικών τωρινών και προηγούμενων εταίρων σας. Λόγου χάρη, η συγκριση Ευρώπη Ευρώπης-Κίνας στη συνεργασία τους με την Αφρική. Διότι ίσως με τους πόρους και τις δράσει μας θα μπορούσαμε να κάνουμε μεγαλύτερη διαφορά. Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε με διαφορετική προσέγγιση Πώς θα μπορούσαν οι δωρητές μας να... Πώς θα μπορούσαμε οι να βοηθήσουμε τα πράγματα. Ναι, πολύ σημαντική ερώτηση και θα ξεκινήσω εγώ. Για τους καινούριου, Κίνα, Ινδία και τους άλλους. Μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι καλή φορείς ως προς την θέση τους παγκοσμίως για τέτοια θέματα. Γι' αυτό όμω χρειάζονται επίσημα να δεξί βοήθεια αναπτυσσόμενε χώρε. Εάν βελτιωθεί το τωρινό σύστημα, θα κάνουν λιγότερη ζημιά εκείνες και οι Ινδίες. Το μόνο που τους μοιάζει είναι το χρήμα και το ψάχνουν με τρόπο απελπισμένο για μια κατασκευαστική εταιρεία στην Ιγυρία, λόγω τάρι, ε, η Κίνα ε, έχει μπει με τα χίλια και αγοράζει άδειε από την Ιγυρία. Στην ουσία κλέβει όμω. Κλέβει χρήμα που πηγαίνει από την Αφρική και την Ιγυρία στην Κίνα. Αυτό το χρήμα δεν πρόκειται ποτέ να μετρηθεί και ποτέ να υπάρξει οποιαδήποτε λογοδοσία. Όμω μπορούμε κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Εάν βελτιώνονταν και ενισχύονταν οι φορολογικές μας αρχές, εάν οι φορείς της διαφθοράς ενισχύονταν, Μπορεί να υπάρξει διαφορά. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η Κίνα και σε πολύ μικρότερο βαθμό η Ινδία. Για να βοηθήσετε, δεν ξέρω αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Ινδία, την Κίνα αποτελεσματικά. Βοηθήστε μας όμως να οπλιστούμε και να τα αντιμετωπίσουμε αυτά που μόνοι μας στη χώρα μας. Ευχαριστούμε. Πολύ σύντομα. Ναι, υπόθηκαν κάποια πράγματα. Όταν ε, ε, μιλάμε για τα θέματα αυτά, η δική μου η αξιολόγηση είναι ότι κάποιες φορές η συζήτηση έχει να κάνει για το σκηνή και το πόσο μακρύ είναι ένα σκηνή με το οποίο τελικά θα σας κρεμάσουν. Δείτε τι έγινε σε χώρε όπως η Σιέρα Λεόν. Βεβαίω η Κίνα τελικά ενδιαφέρεται για τι εταιρείε τη εν τέλει. Αυτό τονίζει την ανάγκη, θυμίζει την ανάγκη για το πόσο χρειαζόμαστε διεθνείς κανόνες που να ισχύουν για ευρωπαϊκές, αμερικάνικέ αλλά και κινέζικες εταιρείε. Είναι δίκαιος ο διαχωρισμός αυτός, ότι χρησιμοποιούν την ίδια κλίμακα οι νέες χώρες για το πώς εκμεταλλεύονται τους πόρους στις διάφορες χώρες της Αφρικής. Όμως μόνο με ένα παγκόσμιο σύστημα μπορούμε να τα ελέγξουμε αυτά. Και χρειάζεται ένα πλαίσιο του ΟΗΕ. Ευχαριστώ. Τέσσερις θέλουν ακόμη, α, πέντε θέλουν ακόμη το λόγο. Ο χρόνος μας ε, θα τελειώσει, θα έχουμε μια σύντομη που είναι κρίθη από τους διερμηνείς, μια σύντομη παράταση. Σας παρακαλώ να γίνουν ε, όλες μαζί ερωτήσεις και να τις απαντήσετε από κοινού. Ανελής είναι η πρώτη. Άρνελής, συγγνώμη. Ευχαριστώ, όπως είπε και η Έλλη Είχαμε ε, πολύ καιρό που το θέλαμε αυτό. Έχουμε τις, ε, τις συνόδους ε, Ευρωπαϊκής, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γνωρίζουν τα Panama Papers και να διερωτώνται τι να κάνουν για όλα αυτά. Δεν ξέραμε για την Κένια και είπαμε ότι θα το θίξουμε γιατί θα έχουμε έκθεση από το Ευρωκοινοβούλιο. Οπότε θα το θίξουμε και πάλι στην σύνοδο της ΑΚΕ, ίσως όχι στην επόμενη αλλά στη μεθεπόμενη. Και πολύ θα ήθελα καρποφόρα εργασία και από τη δική σας πλευρά για να μπει το θέμα και στην ΑΚΕ. Άψογη του χρόνου. Εύα Ζουλή. Σας ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση για το ρήπατο, τον νούχου ρήπατο. Μπορούμε να συμφωνήσουμε για το γεγονός ότι εάν οι ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν εφαρμόσει τους κανόνες ε, τη, το καιρό του Αμπάσα δεν θα είχε μπορέσει να κρύψει δισεκατομμύρια δολάρια. Ε, είδαμε ότι χρησιμοποίησε ευρωπαϊκούς φορολογικούς παραδείσους ή ευρωπαϊκές τράπεζες. Νομίζω 15 χώρες και 43 λογαριασμοί βρέθηκαν τότε. Και ξέρω τον αγώνα που έχει κάνει η Νιγηρία για να πάρει πίσω αυτά τα χρήματα και ποτέ στην πράξη δεν τα πήρε πίσω. Η ερώτησή μου είναι, σήμερα η κυβερνήτες σα, γιατί νομίζω πολλοί από αυτού είναι ακόμα διαφθορημένοι και κλέβουν τα χρήματα, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ευρωπαϊκές τράπεζες ή μετακινήθηκαν σε άλλες χώρες. Η Χάοιντι Χάουταλα. Χαουιντι χαουταλα Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Εγώ όταν ήμουν υπουργό υπεύθυνη για την ε, διεθνή ανάπτυξη είχα και την ευθύνη ε, για την παρακολούθηση και την υποπτία των κρατικών εταιριών. Αν είχα την επεποίθηση λοιπόν ότι αν θέλουμε να εξαρθρώσουμε την, ε, τη διαφθορά υψηλού επίπεδου και φυσικά και γνωρίζουμε τον βασικό ρόλο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας offshore θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς την κρατική ε, να παραμένουν μάλλον κρατικές επιχείρησεις, γιατί πολλές φορές ε, ο πλουτισμός αυτός ορισμένων ανθρώπων είναι, οφείλεται στην ιδιωτικοποίηση κρατικών ε, επιχειρήσεων. Ο ΣΑ έχει συστήσει αυτό, προσπαθεί να αποφύγει συγκρούσεις συμφερόντων, έτσι να δημιουργηθεί η διαφάνεια. Εσείς πιστεύετε ότι εκεί κάτι μπορούμε να ενθαρρύνουμε από την αναπτυξιακή πλευρά για να βελτιώσουμε την οικοδόμηση δυνατοτήτων. Άννα να σας πω πρώτα απ' όλα ε, έχουμε μία μονάδα τώρα στην DG ανάπτυξη, που θέλουμε να βοηθήσουμε έτσι τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης να ανακτήσουν ε, περιουσιακά στοιχεία, όχι μόνο όμως εκείνες αλλά και όλες τις χώρες που το προσπαθούν. Ρωτήσαμε συχνά το ρόλο των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι όλα ένα και περισσότερε ευρωπαϊκέ τράπεζε αγοράζονται από πολύ διεφθαρμένου ανθρώπου, όχι μόνο από αναπτυσσόμενε χώρε. Δείτε για παράδειγμα το ρόλο τη οικογένεια Ντοσάντο ε, τη Αγκόλα στι πορτογαλικέ τράπεζε. Και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ο αντιπρόεδρος της Αγγόλα, ο κύριος Ντο Σάντος, πρόεδρος της Οναγκόλ, ε, καλέθηκε, καλέστηκε στην... Ε, μάλλον, συγγνώμη, ε, είναι σε δίκη στην Πορτογαλία γιατί αγόρασε έναν εισαγγελέα. Και ήταν πολύ υγιής η αντίδραση της πορτογαλικής δικαιοσύνης. Τι κάνει το δικό σας δικαστικό σύστημα, αντιδρά επίσης, είναι Η κυρία Σκοτ Κάτω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξέρω τι πιστεύετε για την ιδέα του Παγκόσμιου Σώματος, Φορολογικού Σώματος του ΟΗΕ. Επίσης, πέρσι στη Λονδίνο έγινε μία ε, σύνοδος για τη διαφάνεια με τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων βουλευτών Θεωρείτε πως αυτό είναι θετικό, ακόμα και οι κυβερνήσεις μας στηρίζουν αυτή την ατζέντα και έπειτα τι πιστεύετε για την ιδέα της συμπερίληψης ρητρών ε, κατά της ε, φοροαποφυγής σε όλες τις συμφωνίες που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Και τώρα Χουάν Φερνάντες ε, Λόπες Αγγιγιάρ, καθηγητά. Η ερώτησή μου ακολουθεί την ίδια γραμμή όπως αυτή τη συναδέλφου Εύα Ζολή και της Άννα Γκόμας. Και σας την απευθύνω σε εσά κύριε Μαζιώμα, που είστε εκπρόσωπος του δικτύου για τη φορολογική δικαιοσύνη στην Αφρική. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για τις δυνατότητες βελτίωσης της στρατηγικής για τους πόρους που κατάσχονται από τους ηγέτες των ε, διεφθαρμένων ορτισόμενων χαρών, για παράδειγμα του πρώτου γιου και προφανώς του κληρονόμου του Προέδρου της σημερινής Γουινέας, το οποίο τα περιουσιακά στοιχεία έχουν κατασχεθεί στη Γαλλία και στην Ισπανία. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε τα κατεσχημένα περιουσιακά στοιχεία ε, ή χρήματα να επανεπενδυθούν ε, στις αναπτυσσόμενες αυτές χώρες. Ευχαριστώ και για την πειθαρχία σας. Τρία λεπτά για τον καθένα από τους δύο ομιλητές μας και κατόπιν θα ολοκληρώσουμε. Παρακαλώ, ξεκινήστε. Και ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Λοιπόν, το βασικό συμπέρασμα που είναι και σαν προμετωπίδα της τελικής έκθεσης του υψηλού επίπεδου ομάδας εργασίας είναι παρακολουθήστε το, σταματήστε το, συλλάβετε το. Αυτά είναι τα τρία βήματα. Να παρακολουθήσετε, δηλαδή να ξέρουμε πώς κινείται το χρήμα. Εδώ είναι κλειδί η διαφάνεια. Τι συστήματα, τι παγκόσμιες δομές βοηθούν την ε, ροή, την παράνομη του χρήματος. Δεύτερον, αφού ξέρουμε πού έχει πάει το χρήμα, τι μπορούμε να κάνουμε για να το σταματήσουμε. Αυτό είναι να υπάρχουν σε όλες τις συμφωνίες ε, ρήτρες κατά τέτοιου τύπου πρακτικές. Υπάρχουν μια σειρά από βήματα που είναι ήδη ε, έχουν θεθεί από διάφορες οργανώσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή, ώστε να κλείσουμε τα παραθυράκια. Και τρίτον, εδώ είναι το κρίσιμο. Όταν βρούμε που είναι τα χρήματα αυτά τελικά που έχουν καταλήξει, πώς θα τα ανακτήσουμε. Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνουμε ότι οι διαδικασίες για την ανάκτηση πόρων είναι τόσο περίπλοκοι Δεν ξέρω αν τα χρήματα του Αμπάτζα με όλες τις προϋποθέσεις που τίθεται στις κυβερνήσεις δεν ξέρω αν τελικά τα έχουμε λάβει. Κοίταξε, μου κλέψε το χρήμα μου. Και όταν πάω να το ξαναπάρω, ε, μου επιβάλλει τόσο περίπλοκου κανόνε που δεν μπορώ να το κάνω. Τώρα για μια παγκόσμια φορολογική αρχή. Ναι, σωστή θα ήταν ε, μια τέτοια πρωτοβουλία. Έχουν γίνει κάποια πρώτα βήματα, δημιουργείται περισσότερη ε, αποδοχή. Υπήρχαν ε, αντιδράσεις, την άντιση ήταν πολύ ψηλότερη από ό,τι σήμερα και νομίζω ότι και το Κοινοβούλιο σας θα μπορούσε να το θέσει ως προτεραιότητα να ενισχύσουμε και από τεχνική και από οικονομική και από πλευρά προσωπικού αυτή την επιτροπή που υπάρχει ήδη για τα φορολογικά θέματα και να διευρύνουμε την εντολή της. Και συμφωνώ με τον ρόλο των βουλευτών. Και προσωπικά βεβαίω. Βλέπουμε παραδείγματα σε πολλές αφρικανικές χώρες, Κοινοβουλευτικοί θέτουν αυτά τα θέματα και ε, έχουν και την αναγκαία γνώση για να θέσουν τις σωστές ερωτήσει γιατί πολλές φορές πολλές φορές είναι δύσκολο να εκθέσεις αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δημιουργούν τα αναγκαία δίκτυα για να μαθαίνουν οι μένα από τους δε, να ε, ανταλλάσσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Και τέλος, για το θέμα της εταιρική διακυβέρνησης. Συμφωνώ. Παρατηρούμε μια τάση αυξάνονται ε, οι διαδικασίες ε, ιδιωτικοποίησης. Τα κράτη επιχειρούν να ε, συμμετέχουν λιγότερο στην οικονομία. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν έχει τεθεί ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο. Να, να ε, διαχειριστούμε δηλαδή σωστά αυτή τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ριμπαντού. Πολύ γρήγορα. Ναι, έχουν γίνει πολλές αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα. Χάρη εν μερικές τις δικές σας αλλαγές για τους δικηγόρους, τις επιχειρήσεις υλοποιούνται καλύτερα και περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Βεβαίως, υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις όπου οι διεφθαρμένοι της Αφρικής κρύβουν το χρήμα τους σε περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη. Πάντως, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου συνέλαβαν, λέει, τον πρώην Υπουργό Πετρελαίου της Νιγηρίας και δεν είναι ο μόνος. Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται. Φεύγει τόσο χρήμα από την Αφρική και το επενδύουν σε ιδιοκτησία στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η αλλαγή. Απαντήσατε στην ε, κυρία από τη Φιλανδία, μια χαρά. Σας Ευχαριστώ και σας πολύ. Δεν ήξερα ότι είστε εσείς οι ίδια. Σας ευχαριστώ γιατί μας έχετε βοηθήσει φοβερά. και το θέμα της ανάκτησης των της χρήσης μάλλον των πόρων που έχουν ανακτηθεί. Πήραμε, όπως σας έλεγα, ένα δις δολάρια κάποια στιγμή από ένα ελβετικό λογαριασμό. Εκείνη τη στιγμή ε, οι ελβετικές αρχές επέμειναν ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ευθύ αμέσω οι πόροι αυτοί σε πράγματα χειροπιαστά, υπαρκτά για τους πολίτες. Και τελικά το κάναμε και δεν το μετανιώσαμε, διότι κάποιοι πήραν αυτό το χρήμα από εμάς, μας το πήραν, το πήγαν σε άλλη δικαιοδοσία. Και τελικά δεν είναι λάθος να επιμένει κανείς το χρήμα αυτό να χρησιμοποιηθεί νομίμως. Ένα μεγάλο σχολείο, ένα μεγάλο νοσοκομείο. Πάρτε το χρήμα, είπαμε, Χρησιμοποιήστε το για να χτίσετε ένα κτίριο παραπάνω. Είναι ένα μήνυμα κι αυτό. Εγώ ήμουν επικεφαλής της Νιγηρίας που συζητούσε αυτά τα θέματα στο επίπεδο του ΙΕ και η Ελβετία τα επέστρεψε τα λεφτά και τα χρησιμοποίησαμε ακριβώς για κοινωνικά έργα. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς πώς. Είναι να παίρνει κανείς το χρήμα και να φροντίζει από αυτό να έχει κάποια χρησιμότητα. Για να μην σπαταλιέται τελείω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο μιλητές θερμότατα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων, θαυμάσια ακρόαση. Μάθαμε πολλά για τις προσπάθειες που γίνονται στην Αφρική και μέσω της διεθνούς συνεργασίας και μέσω του ρόλου της Ευρώπης για να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Φιτς Γκίμπον, το οποίο το μήνυμα θα βάλουμε στο, στον ιστοτόπο μας. Ευχαριστώ και για τις γραπτές απαντήσεις που μας υποβάλατε και σας παρακαλούμε. Αν έχουμε επιπλέον ερωτήσεις ε, θα μπορούσαμε να σας τις στείλουμε γραπτά για να μας δώσετε απαντήσεις. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τους διερμηνείς. Και όπως είχαμε πει, όπως είχαμε αποφασίσει και συμφωνήσει να την κλείσω ε, μετά τα 10 του παράταση που είχε ε, συμφωνηθεί. Okay.